Welcome to everybody. You can take the, your seat, please. Καλώς ήλθατε, αν θέλετε να καθίσετε. Και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, λέει η Πρόεδρος και συνεχίζω στα Ιταλικά. Να καλωσορίσω τους φιλοξενουμένους, τους εμπειρογνώμονες που έχουμε μαζί μας σήμερα για ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο αυτό που συζητούμε σήμερα για την λαθρεμπορία και καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς ε, μεταξύ άλλων και στο Ιράκ θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ταχύτατα αν μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερησίας διατάξεως, όπως και το σχέδιο πρακτικών της προηγουμένης συναντήσεως. Αν δεν έχουμε κάποιες αντιρρήσεις, θα θεωρήσω ότι αυτά τα δύο είναι εγκεκριμένα. Ζητώ συγγνώμη. Πολύ σύντομα ένα σχόλιο σχετικά με τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Σχετικά με το φόρουμ της διαδικτυακής διακυβέρνησης έχει γίνει μια σύγχυση με το ε, διοικητικό φόρουμ. Δεν υπάρχει όμως κανένα διαδικτυακό φόρουμ για τη διοίκηση. Παρακαλώ να διορθωθεί. Σεντσάλτρο. Οπωσδήποτε, έχετε δίκιο. Και με την διευκρίνηση αυτή μπορούμε να περάσουμε σημείο Τρία λέει πρόεδρος. Σήμερα έχουμε κάλυψη με διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Καλησπέρα σας και από την ελληνική διερμηνία. Ε, έχουμε και web streaming καταγραφή της σημερινής ε, συνεδριάσεως. Και να πω ότι μεταξύ των εγγράφων σήμερα θα βρείτε και μια σύντομη έκθεση επί της ε, πρόσφατης αποστολής ε, στην αφιπολη 16 16-19 Ιουνίου στην Ελλάδα και καθότι ηγούμενη της αποστολής μου φαίνεται ενδιαφέρουσα σύμπτωση που σήμερα ενημερωνόμαστε σχετικά με αυτό γιατί όπως γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι που ήταν μαζί με εμάς στη σημαντική αυτή επίσκεψη Νομίζω ότι πληρώσαμε τα καθήκοντά μας με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε, διότι οι βασικές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα πρέπει να συνυπολογιστούν με πολλά ακόμα θέματα και νομίζω ότι η συμφωνία στην οποία φτάσαμε σήμερα μετά από πολύ κόπο και που ίσως ελπίζουμε προσφέρει μία έστω και οδυνηρή δυνατότητα για τον ελληνικό λαό και για την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να πω επ' αυτού ότι ξεπεράσαμε ένα δύσκολο πέρασμα, εγχείρημα που διακύβευε το μέλλον του ελληνικού λαού και της Ευρώπης. Ήθελα απλώς να πω όν passant». Τώρα, προτού παρουσιάσω τους τέσσερις ε, εμπειρογνώμονες που έχουμε σήμερα μαζί μας, θα ήθελα να πω κάποια ολίγα. Η Κομισιόν εκπροσωπείται εδώ μαζί μας, ε, όπως και το Συμβούλιο, γιατί θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική δράση. Όλοι έχουμε κατά νου τους ε, πολεμιστές της ISIS που καταστρέφουν διάφορα κοιμήλια της πολιτιστικής παράδοσης χειρόγραφα παλαιά στο Ιράκ λοιπά, Αγάλματα και ούτω καθεξής κτίρια. Μιλάμε για ε, τα αγάλματα του Βούδα στο Μπαμιάν, ε, στο Ρούτ, στο Τιμπουκτού, στην Παλμύρα όπου είχαμε καταστροφές αλλά και 300 άτομα που προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα κοιμήλια αυτά ε, Είμαστε ενώπιον μιας τραγωδίας και ανθρώπινης και πολιτιστικής. Έχουμε 10.000 πρόσφυγες μόνο στην ε, Συρία. Έχουμε μια τραγική κατάσταση η οποία βλέπει 50.000 να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τη χώρα τους και να προσπαθούν να σωθούν και έχουμε και μια συνειφασμένη κατάσταση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητος και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως ε, στο Κοινοβούλιο με το ψήφισμα μαζί με την Επιτροπή ε, Πολιτιστικών Θεμάτων συζητήσαμε την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από της Κομισιόν και Συμβουλίου γνωρίζουμε βέβαια τα κενά που υπάρχουν εδώ και τις ελλείψεις αλλά είπαμε ότι όταν φωνεύονται άνθρωποι και παραβιάζονται τα θεμελιώδη συστατικά και στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξής μας και καταστρέφουμε στοιχεία της πολιτιστικής μας κοινή παράδοσης και κληρονομιάς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το θυμάστε τον Απρίλιο στο ψήφισμά μας ότι είχαμε αναλάβει δέσμευση όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Ε, έχουμε και εκπρόσωπο τη UNESCO εδώ στις Βρυξέλλε, την Ναμπουκόβα, η οποία, με την οποία θα συζητήσουμε και το Σεπτέμβριο ε, επί άλλου θέματος και συνημεριζόμαστε και την εκστρατεία ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου εκ μέρου των ΗΠΑ από αυτού το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ επίσης σχετικά με τις παράνομες πωλήσει που προέρχονται από Συρία και Ιράκ τέτοιων στοιχείων πολιτικής κληρονομιάς. Έχουμε κάποια μέσα προστασίας, έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τον πλούτο αυτόν. Έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε και να αναστηλώσουμε και να ανακαινήσουμε στο μέτρο δυνατού όλα αυτά τα κοιμήλια. Έχουμε ψηφίσματα και αποφάσεις της UNESCO σχετικά με τις παράνομες εξαγωγές και διαθέσεις ε, στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, περιουσιακών στοιχείων δηλαδή πολιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή τράπεζα δεδομένων πολιτισμικών ε, στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και άλλων. Έχουμε την ε, βάση δεδομένων Λεωνάρντο που κατέγραψε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τέτοια στοιχεία υπό τις ε, Ιταλικές Αστυνομικές Αρχές. Χρειαζόμαστε όμως τη συνεργασία όλων. Είχαμε και ένα συνέδριο της ε, Μεσογειακής Συνδιάσκεψης στη Ραμπάτ που ολοκλήρωσε τις εργασίε της ε, με δέσμευση μεγαλύτερης και αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων και των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, ώστε να έχουμε ένα σχέδιο δράσεως προκειμένου να ενσωματώσουμε, να οργανώσουμε καλύτερα όλες αυτές τις προσπάθειες. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται ως ηγέτης με τις οδηγίες και τις νομοθεσίες της σχετικά με την παράνομη διάθεση κοιμηλίων της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και εξάλλου το είχε πει και η Κομισιόν αυτό κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος ή στην Ολομέλεια ότι γίνεται και μια μελέτη ώστε να στοχευθεί μια οδηγία επί των της εισαγωγής γιατί σε αυτό έχουμε συγκεκριμένες ελλείψεις τέτοιων λοιπόν στοιχείων και πρέπει να υποστηρίξουμε την ευαισθητοποίηση, την ε, προσπάθεια εκπαίδευσης όλων απέναντι στην αξία αυτών των κοιμηλίων, Μιλάω για σπουδαστέ, μιλάω για ακαδημαϊκούς, μιλάω για ερευνητές, μιλάω για ανθρώπους που εθελοντικά συμμετέχουν στη Συρία στο πεδίο για να υπερασπιστούν τα κοιμηλία αυτά. Πρέπει λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε τα οικιανόκρινη να αυξήσουν την ακτίνα δράσεώς τους προστασίας των κοιμήλιων αυτών. Υπάρχει και μια χάρτα που πρόσφατα ενεκρίθη σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με ε, ε, φυσικές καταστροφές, εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο ακριβώς παρέμβασης επί στοιχείων πολιτικής κληρονομιά αντίστοιχα με άλλα ακίνητα στοιχεία περιουσιακά. Και εδώ μιλούμε για εγκλήματα, εγκληματικές δράσεις που ε, γίνονται τακτικά και γίνονται και με μία, αν θέλετε, πρόθεση πολιτιστικής εκαθάρισης Επομένως δεν πρόκειται μόνο για έγκλημα πολέμου, αλλά όπως είπαμε στο ψήφισμα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, εδώ έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος με τις δράσεις αυτές, τις πράξεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ηγείται παγκοσμίω, είναι ο πρώτος υποστηρικτής ε, της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής πλειονομιάς, για την αναστήλωση, για την ψηφιοποίηση της καταγραφής των στοιχείων αυτών, αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά, πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Στην ευαισθητοποίηση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα, της ε, συλλογής ε, πληροφοριών, της συνεργασίας με την Interpol, η οποία δουλεύει πολύ στον τομέα αυτόν. Και οπωσδήποτε τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ε, συνομιλητές μας, διευκρινίζοντας όμως ότι όπως είδατε αποφασίσαμε από κοινού με την Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς να διακρίνουμε σε δύο πάνελ τη συνάντησή μας τη σημαίνει. καταρχάς επί της καταστροφής και πολιτιστικής κληρονομιάς σχετικά με αυτά που πρέπει να γίνουν λοιπόν για την αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού και δεύτερον για τη λαθρεμπορία το μαύρο εμπόριο αυτών των στοιχείων. Και στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε και ένα βίντεο ένα μικρό βίντεο, εμπαστητώσει, ως μαρτυρία. Θεωρούσαμε αξιόλογο και σημαντικό. Του καθηγητού Αμούν Αμπτούλ Καρίμ από το Μουσείο Πολιτικής Κοινωνίας Συρίας, όπου 25 Οκτωβρίου του 2014 έλαβε ένα βραβείο προστασίας παγκόσμιας πολιτικής κοινωνίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη δουλειά του σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την προστασία ακριβώς της ρακινή Πολιτική κοινωνία. Τώρα θα έδινα το λόγο λοιπόν, παρουσιάζοντα του ε, συμπαρουσιαστέ του πάνελ, ε, ξεκινώντα από τον καθηγητή Λαντζερίνη, από το Μεσίνιο Σιένα, στο διεθνέ Δίκαιο τη προστασία ε, των Κυμελίων τη Πολιτιστικής Κληρονομία, θα μα δείξει πώ τα τρίτα κράτη και οι διεθνεί οργανισμοί μπορούν να παρέμβουν προ την προστασία των κυμελίων αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, μαζί με την ευθύνη και την αρμοδιότητα της προστασίας. Ε, θα ήθελα όλοι, παρακαλώ όλους, να σεβαστούν τα 8 λεπτά. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη θυσία από μέρους σας, αλλά έτσι θα έχουμε χρόνο για όλους. Παρακαλώ κύριε Λαντζερίνη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτιστικής Κοινωνίας γιατί είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας Κυρία ήδη σα έκανε μία εισαγωγή του τι θα ακολουθήσει την παρουσίασή μου και ελπίζω να έχετε δει τι εικόνε. και να είστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει, τι γίνεται ακριβώς. Τώρα, με νομικού όρου. μπορώ να σας πω ότι η καταστροφή πολιτισμικής κληρονομιάς, όταν γίνεται εσκεμένα και δεν συνδέεται με κάποια στρατιωτική ανάγκη, θεωρείται σήμερα ε, διεθνές έγκλημα. Η κυρία Κώστα τόνισε ότι εκτός από αυτό θεωρείται και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο παρελθόν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έγκλημα δίωξης, διότι ο στόχος δεν είναι η ίδια η πολιτισμική κληρονομιά. Στόχος είναι οι άνθρωποι, οι κοινότητες οι οποίες φαίνονται μέσα από αυτήν την πολιτισμική τους κληρονομιά. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι η καταστροφή της πολιτισμικής ταυτότητας των κοινοτήτων αυτών. Επίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς θεωρείται ε, συστατικό στοιχείο της πρόθεσης για γενοκτονία κάτι που έχει εγκριθεί και τονιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, η κυρία Κώστα αναφέρθηκε στο πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με αυτό, η καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελεί απειλή στην παγκόσμια ασφάλεια, δηλαδή εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, θεωρώντας την, την ε, καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς έγκλημα, υπάρχει και η ευθύνη προστασίας των ε, πολιτών και της ε, πολιτισμικής κληρονομιάς. Και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ευθύνη προστασίας βρίσκεται στο κράτος το οποίο λαμβάνει η χώρα. Όμως όταν το κράτος αυτό είτε δεν είναι σε θέση είτε δεν επιθυμεί την προστασία της ε, πόλης, της κληρονομιάς και του πληθυσμού από αυτήν την ασκεμένη πράξη, τότε υπάρχει μια συλλογική ευθύνη προστασίας, συλλογική ευθύνη της ε, διεθνούς κοινότητας. Συγκεκριμένα η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να βοηθήσει το εν λόγω κράτος και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να γίνει πρόληψη και να αποτραπεί η καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς. Τώρα, η ευθύνη προστασίας. Τι περιέχει. Περιέχει τρεις περιπτώσεις. Καταρχάς, η ευθύνη της πρόληψης. Έπειτα, η ευθύνη της αντίδρασης και η ευθύνη αναδόμησης. Βέβαια, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καταστροφής πολιτισμικής κληρονομιάς μιλάμε για την καταστροφή που λαμβάνει η χώρα από την ε, ίσης. Είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε, στη συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση, όμως δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν σε όλο τον κόσμο και στόχος μας είναι να βρεθεί μια σταθερή μακροπροθεσμή λύση. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι καταρχάς υπάρχει η ευθύνη αντίδραση σε αυτήν την πράξη καταστροφής η οποία έχει διαπραχθεί στα εδάφη τα οποία κατέχει η ίσης. Μπορούμε επίσης να, να θεωρήσουμε ότι μόνο τα διπλωματικά μέσα δεν θα είναι σε θέση να σταματήσουν από μόνα τους αυτήν την ε, καταστροφή, αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Η μόνη πιθανή λύση δυστυχώς είναι η στρατιωτική παρέμβαση, η οποία υπό το διεθνές δίκαιο είναι θεμητή εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλεία. Το Συμβούλιο λοιπόν Ασφαλείας έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει μια στρατιωτική παρέμβαση και ο ρόλος επομένως των διεθνών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου και των κρατών μελών είναι να ασκήσουν πίεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έτσι ώστε να πιστεί για την λήψη μιας τέτοιας λεπτής απόφασης. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτύχει στο να αναλάβει τις υποχρεώσεις του, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τέτοια μέτρα. τα οποία προβλέπονται και από το ψήφισμα 377 του 1950. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση που θεωρώ αρκετά σημαντική. Γνωρίζουμε ότι η ίσης επιθυμεί να επεκταθεί, να επεκτείνει την κατοχή της, όχι μόνο στις, ε, γύρω, στα γύρω εδάφη, όμως και σε άλλα εδάφη. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αίγυπτο, στην Τινησία. Είναι επομένω πάρα πολύ σημαντικό οι διεθνεί οργανισμοί, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δράσουν έτσι ώστε να προληφθεί κάτι τέτοιο, να ε, αποτραπεί αυτό που συνέβη στη Συρία, στο Ιράκ και τη Λιβύη να επαναληφθεί και σε άλλα εδάφη. Και πιστεύω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όταν ε, γίνεται λόγος για πρόληψη. Δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτική δράση. Υπάρχουν πολλά μέτρα που μπορούν να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προληφθούν περαιτέρω καταστροφικές ε, πράξεις. αυτά τα μέτρα μπορούν να είναι, για παράδειγμα, διάφορες πρωτοβουλίες, ευαισθητοποίηση του κοινού, των μέσων ενημέρωσης, ενημέρωση των, ε, της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών, των εγχώνων κοινωνιών, ενημέρωση του λαού για την σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς. Επίσης, καταρτισμός εμπειρογνωμόνων, καταρτισμός στρατιωτικού προσωπικού, ε, κατάρτιση, με συγχωρείτε, ε, ε, της αστυνομίας. Έγκαιρη ενημέρωση. Στήριξη από διεθνή δικαστικά σώματα, για παράδειγμα το Διεθνές Δικαστήριο. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να δικαστούν όσοι καταστρέφουν πολιτισμική κληρονομιά. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η βελτίωση και η αύξηση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα την UNESCO, αλλά και διάφορους τοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα εδάφη που λαμβάνει η χώρα η καταστροφή. Επίσης, πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να αποτραπεί ο επανοπλισμός της ε, ίσης. για να μην επαναληφθούν ξανά αυτές οι καταστροφές. Πολλά μέτρα επομένω μπορούν να γίνουν. έτσι ώστε να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον ε, καθηγητή Λεντζερίνη που μας θύμισε την πολύ σημαντική, την πολύ σοβαρή αυτή ευθύνη και πολύ επίγουσα αυτή ευθύνη την οποία αισθανόμαστε μαζί με, τις, με τους περιορισμούς μας. Γιατί βεβαίως δεν είναι συντονισμένοι, εναρμονισμένοι όλοι οι φορείς ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως θα έχουμε και συζήτηση από αυτού τώρα. Και μετά τις παρεμβάσεις σας βεβαίως θα δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα έδινα τώρα το λόγο στον καθηγητή Ντεκάρο από το International Center for the Study of Cultural Property βάστος από το Διεθνές Κέντρο του Μελετών για την Πολιτική Κληρονομιά και σχετικά με την ενημέρωση των διαφόρων φορέων και οργανισμών ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Θα μας εξηγήσει λοιπόν ο καθηγητής πώς μπορούν να δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί αυτοί καλύτερα και ποιες είναι οι δεσμεύσεις που μπορούμε να λάβουμε. Σας ευχαριστώ για την ε, προσκλησή σας. Θα μιλήσω στα Ιταλικά διότι θα είμαι πιο αποτελεσματικός έτσι. Τι είναι λοιπόν η ICROM. Πρόκειται για μια διακυβερνητική οργάνωση. Σε αντίθεση με την ICOMOS και την ICOM που είναι επαγγελματική φορείς, εδώ εκπροσωπούνται κυβερνήσεις. Υπό την έννοια αυτή είναι ένας πολιτικός φορέας. 134 κράτη εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή. Εκπροσωπούνται. Το 56 δημιουργήθηκε από την UNESCO με ψήφισμα ώστε να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος από την UNESCO φορέας, ο οποίος όμως θα δρούσε εντός των ορίων της εντολής της UNESCO. Τεχνικός φορέας λοιπόν για τους ειδικού και εμπειρογνώμονες στην ε, συντήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής συνομιλία. Έχει έδρα ή στην Ιταλία από το 1958 και από πέρυσι έχει περιφερειακή έδρα ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στην Σάρτζα με αποστολή που αφορά στις αραβικές χώρες. Αυτό είναι σημαντικό για, την, ε, για τις δυνατότητες δράσεως που έχουμε Στι ενεχόμενες χώρες. Πρόκειται για έναν οργανισμό που έχει διαδραματίσει σημαντική, ε, σημαντικό ρόλο σε τοπικά και περιφερειακά προγράμματα. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν εκείνο για την Αφρική. Δηλαδή την σχολή της πολιτιστικής κληρονομίας της Αφρικής. Ένα ταμείο που είχε δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια και που διαχειρίζεται η Ίκρομ που αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την Παναφρικανική Ένωση ως οργανισμό φορέα με παναφρικανική αξία, με έδρα στην Μπενίν. Συνίσταται λοιπόν από τις συνεισφορές, μάλλον υποστηρίζεται από τις συνεισφορές ε, προς τα Ηνωμένα και την UNESCO όλων των κρατών μελών και κατά 30% έχει χρηματοδότηση ε, πέραν του τακτικού προϋπολογισμού. Κάθε δύο χρόνια συνέχεται η Ολομέλεια με Διοικητικό Συμβούλιο 25 ειδικών επαγγελματιών από τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου. Έχει μια δομή επιχειρησιακή πάρα πολύ μικρή, 34 άτομα αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων 14 επαγγελματίες, μια ελαφριά δομή και το οποίο αναγκάζει και αυτό είναι το σημαντικό, σε συνεργασία. Κανείς δεν μπορεί να είναι εμπειρογνώμων επί των πάντων. Συνεργαζόμαστε με τα κέντρα, τα πανεπιστήμια, τους ακαδημαϊκούς φορείς παγκοσμίω που έχουν τις καλύτερες ε, ειδικεύσει ή στην προστασία της πολιτικής ε, κληρονομιάς και για τη συντήρηση και για την αποτροπή κινδύνων και απειλών διαιρούμεθα αυτή τη στιγμή σε τρεις τομείς, επικοινωνία, σημαντικό, ε, ακίνητα στοιχεία πολιτικής ε, κληρονομιάς και κινητά. Επόμενος, συνεισφέρουμε στην συντήρηση και την αποκατάσταση της πολιτικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, αναπτύσσοντας ε, και υποστηρίζοντας όλες τις συνθήκες που διευκολύνουν την προστασία αυτή, τη λειτουργία αυτή. Μιλούσαμε λοιπόν για τεχνική βοήθεια, για την χρηματοδότηση μελετών συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά η ανάπτυξη της κοινότητος που επιθυμεί την προστασία του πολιτισμού αυτού. Επομένως, πέρα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μιλούμε πλέον για την ανάπτυξη δυναμικού, δηλαδή την ανάπτυξη μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας, η οποία θα είναι ικανή να προβαίνει σε αυτήν τη συντήρηση και αποκατάσταση. Κάτι που βλέπουμε στα πλαίσια της κρίσης αυτής είναι ότι πολλοί από τους ε, εθελοντές πολεμιστές ε, που κατευθύνονται προς τη Συρία, το Ιράκ κτλ. προέρχονται από δυτικές αν όχι ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο δημιουργεί το εξή πρόβλημα. Μας δείχνει μια έλλειψη, ένα κενό στο εκπαιδευτικό σύστημά μας ή το σύστημα ανάπτυξης δυναμικού, διότι δεν υπήρξαμε ικανοί τις τελευταίες δεκαετίες, ήμασταν μεν ικανοί να αναπτύξουμε τεχνικές δεξιότητες, αλλά όχι να αναπτύξουμε κοινωνίες εντός των οποίων οι μετανάστες, οι φτωχοί, οι περιθωριοποιημένοι θα αισθάνονταν ότι η πολιτική κληρονομιά δεν είναι κάτι που αφιερώνεται μόνο για τους ε, υπερπλούσιους στα μουσεία, αλλά κάτι που θα τους ενσωμάτωνε και θα τους ενέτασε στην ευρύτερη κοινωνία. Μια παγκόσμια αποκληρονομιά. Αυτές οι έννοιες όπως και η έννοια του εγκλήματος της ανθρωπότητας έχει σχέση με την ικανότητα του να αισθανθεί κανείς μέλος της κοινωνίας. Επομένως τα εγκλήματα όπως στην Μόζουλ μεταξύ άλλων στο μουσείο δεν είχαμε ομοιογενή αντίδραση από πλευρά τη διεθνή κοινότητα. Γιατί όταν κάποιο καταστρέφει κάτι, το κάνει εξ ονόματο ενό τμήματο κοινωνία κατά ενό άλλου τμήματο κοινωνία που είναι ακριβώς το αντίστροφο από την έννοια της ενωμένης ανθρωπότητος ως συνειδιοκτήτης, συνειδιοκτήτριας του στοιχείου αυτού. Σήμερα λοιπόν η εκπαίδευση είναι το α και το ω της κατάρτισης και εκπαίδευσης. Δεν είναι πλέον ο τεχνικός, ο χημικός ή ο αρχαιολόγος με την αυστηρά τεχνική έννοια. Ο ενδιαφερόμενος φορέας, ο stakeholder για το πούμε στα ελληνικά, είναι ο ενδιαφερόμενος στην πτυχή της πολιτισμικής κληρονομιάς και όχι μόνο του τεχνικού, της τεχνικής αξίας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακηρύξεις, αλλά πέραν από την πολιτική τους πτυχή, οι διακηρύξεις αυτές, οι ανακοινώσεις αυτές, επιτρέπουν να φτάσουμε σε μια κοινή αναγνώριση σχετικά με την Αρβική Λίγκα, τους ε, συναρμοδίους υπουργούς ε, παιδείας ε, στη Σάρτζ, η κυρία Μογκερίνη μετά την Παλμύρα, διάφορες δηλώσεις, η κυρία Μπόκοβα της UNESCO, όλες αυτές οι διακηρύξεις ήταν θεμελιώδους αξίας. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και ορισμένα πολύ συγκεκριμένα και αυτά. Όπως το παρατηρητήριο επί της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται από, την UNESCO ε, με, την, με την Ίκρο, και τα λοιπά και άλλους. Άλλη πρωτοβουλία, Άσορ, για τις ανατολικές σπουδέ μαζί με τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το Getty Conservation Institute και το παγκόσμιο, ε, το World Monument Fund, εν πάση περιπτώσει, το Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ για την συνεργασία των Ινστιτούτων για τη συντήρηση της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς ε, του Πανεπιστημίου του Yale. Η Γερμανία με το Syrian Heritage Archive Project, ώστε να καταγράφεται η πολιτιστική αυτή κληρονομιά και άλλες πολλές πρωτοβουλίες. Υπάρχει ένα έργο, ένα πρόγραμμα της UNESCO μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χρηματοδότησε δηλαδή πρόγραμμα της UNESCO, safeguarding of the Syrian heritage στο εσωτερικό του οποίου, στο πλαίσιο του οποίου υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις που και εμείς συμμετέχουμε ως ίκρο και μία από τις εμβληματικές ενέργειες στο πλαίσιο αυτό ήταν ε, οι ομάδες αν θέλετε άμεσου δράσεως μετά από καταστροφές είτε φυσικές είτε ανθρώπινες δηλαδή κατόπιν ενός πολέμου, μιας πολεμικής σειράξεως. Είχαμε λοιπόν μια, ένα πρόγραμμα κατάρτισης στην Ιταλία προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές. Προκειμένου να οδηγήσουμε μια χιονοστιβάδα ε, καθόδου μεταφορά τη γνώσης αυτής. Εδώ ο κύριος που βλέπετε ο Σαλάχα Αιγύπτιος εκπαιδεύτηκε και με τη σειρά του εκπαίδευσε μια ομάδα εκπαιδευτών οι οποίοι τελικά ευρέθησαν στο Κάιρο τη στιγμή που εξεράγει το παγεδεμένο αυτοκίνητο απέναντι στο αστυνομικό τμήμα και το μουσείο της ε, Ισλαμικής τέχνης το οποίο οδήγησε τους Αιγυπτίους να δημιουργήσουν και άλλες τέτοιες ομάδες στο έδαφος. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν να εκπαιδεύουμε τέτοιες ομάδες αμέσου δράσεως, αμέσου βοηθείας σε συνεργασία με τους ωραϊκούς φορείς αυτό το είχαμε κάνει και τον Ιούνιο ή στην ε, Βηρητό για τους ε, δημοσίους υπαλλήλου της ε, Συρίας και εδώ είναι τα υπόλοιμα που, που κάνουμε για την Ιεμένη, την Ισία, τη Λιβύη κτλ. Αυτό που ήθελα να θυμίσω, καθότι αυτό συνδέεται και με την δράση που ανέλαβε ένα λεπτό έχετε, του λέει η πρόεδρος εκτός μικροφώνου του ομιλητή, αυτό, εν πάση το νομοθέτημα αυτό, του, ε, της Αμερικανικής, ε, του Αμερικανικού Κογκρέσου δημιούργησε ένα νέο φορέα που συντονίζει όλες τις δράσεις της Αμερικανικής Κυβερνήσεως σε περιπτώσεις ε, καταστροφών και κρίσεως και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να άρει τους περιορισμούς εισαγών προκειμένου να επιτρέψει safe haven, ασφαλείς λιμένες εισαγωγών στοιχείων πολιτιστική κληρονομιά στι ΗΠΑ. Αυτό το είχε κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε τροποποιήσει με τη σειρά τη την ε, νομοθεσία, την ειδική νομοθεσία που είχε ε, εγκριθεί μετά τις κυρώσει επί της Συρίας, τροποποιώντας μία από τι διατάξει ε, των ΗΠΑ Εθνών, ακριβώς για να επιτραπούν εισαγωγέ σε περιπτώσει κρίσεως, εκτάκτου ανάγκη. Άρα λοιπόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε οργανώσεις όπως η ECOM και η κόκκινη κατάλογή της που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν. Γιατί πρέπει να έχουμε μια τυπολογική καταγραφή των στοιχείων αυτών, των αντικειμένων αυτών που πρέπει να προστατευτούν. Και κάτι τελευταίο. Μακροπρόθεσμα. Όπως βλέπετε εδώ από τα μεγέθη, έχουμε 11 εκατομμύρια πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 4 εκατομμύρια στις άμεσα γειτονικές χώρες, μόνο από την κατάσταση στη Συρία. Δεν μιλάω για τη Λιβύη ούτε τίποτε άλλο. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγοι, τα παιδιά, τα στρατόπεδα, χρειάζονται φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα κτλ. Αλλά είναι προς το συμφέρον όλης της ανθρωπότητας να προσδώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο μια κοινή αξία πολιτιστικής ε, παράδοσης και κληρονομιάς παγκόσμιας αλλά και των ίδιων των χωριών τους, της χώρας τους, της ταυτότητάς τους οι Ευρωπαίοι εφήβραμε τα οικομουσία, τα μουσεία δηλαδή που συνίστανται σε φωτογραφίες, αποτελούνται από φωτογραφίες και εικόνες από το σπίτι μας, το, τον τόπο από τον οποίο προερχόμαστε, για να έχουμε μια επανασύνδεση με τον τόπο αυτόν και να καταλαβαίνει καλύτερα και αυτός που τις υποδέχεται από πού έρχονται, διότι έτσι γεφυρώνουμε εκείνο το χάσμα που οδηγεί στην περιθωριοποίηση. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, λέει η Πρόεδρος, ή ε, στον οποίο ε, δώσαμε κάποια λεπτά παραπάνω γιατί ήταν κρίμα να τον διακόψουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσουμε και θυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε και ένα σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, εκπαίδευση υποσυνθήκες ε, εκτάκτου ανάγκης και αυτή η θεματική ήταν πολύ σημαντική. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζιλ Τζουτέχτχο, που είναι επικεφαλής ε, νομικός εμπειρογνώμονας ε, του, ποινικού, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έχουμε συνεργαστεί σχετικά και με τον καταστατικό κανονισμό του Διεθνούς Δικαστηρίου και έχουμε πάρα πολλές παραπομπές σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σε άλλα πεδία της αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Θα μας δείξετε λοιπόν, θα μας παρουσιάσετε κάποιες ε, πιθανές, ε, πιθανότητες, δυνατότητες παρέμβασης του δικαστηρίου στα παιδιά αυτά και θα μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα κατά πόσον η δική μας ιδέα, το δικό μας σκεπτικό ότι τα εγκλήματα τα ανθρωπότητα συνίστανται, έχουν νομική εξήγηση και μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω και θα είμαι και πολύ συγκεκριμένος. Υπάρχουν ε, συνέπειες μακροπρόθεσμες ε, όταν ε, μιλάμε για καταστροφή πολιτιστικών μνημείων και θα αναφερθώ εδώ σε αυτό που είπε η Γενική Διευθύντρια της UNESCO. Ο πολιτισμός βρίσκεται πολλές φορές στο επίκεντρο κάποιων συγκρούσεων και σειράξεων και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά σαν ένα θέμα ε, ασφάλειας. Τι κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτά τα μνημεία και αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Οι απαντήσεις βεβαίως είναι πολλές, αλλά υπάρχει και η νομική απάντηση. Γι' αυτό και ο ρόλος του ποινικού δικαστηρίου, της ε, δικής μου δηλαδή δικαιοδοσίας, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και όσον αφορά αν θέλετε, τη νομική πτυχή, αλλά και δεν νομίζω θα σας εκπλήξει αυτό που σας λέω. Εδώ και χρόνια, ακριβώς επειδή αυτή η στρατηγική και η πολιτική καταστροφής πολιτικής κληρονομιάς συνίσταται σαν ένα από τα στοιχεία των υποθέσεων που απασχολούν ε, τους εισαγγελείς ε, του δικαστηρίου μας. Είναι κάτι που μας ανησυχεί και θα ήθελα να πω ότι η καταστροφή πολιτικών ε, μνημείων ε, και αγαθών συμπεριλαμβάνεται στο καταστατικό της Ρώμης. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να διωχθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα και πρέπει πραγματικά η διεθνής κοινότητα να εκφράσει τη σημασία που έχουν ε, αυτές οι προσφυγές. Φυσικά και η εντολή του δικαστηρίου είναι να δράσει από κοινού με τους θεσμούς και με τα κράτη. Και εξ ονόματος της ε, εισαγγελέως της κυρίας Σουντά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχουμε σήμερα σε, αυτά, ε, σε αυτήν την συνεδρίαση. Όσον αφορά λοιπόν τη δράση του Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναφερθώ, όπως σας είπα, στο καταστατικό της Ρώμης, όπου μέσω αυτού του καταστατικού διαθέτουμε όπλα και δυνατότητες να προστατεύσουμε την πολιτιστική κοινωνία. Βάσει του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, επίσης βάσει του άρθρου 7 και η καταστροφή των πολιτών αγαθών είναι κάτι που έχει και άμεση σχέση με το έγκλημα της γενοκτονίας που επίσης αναφέρεται στο καταστατικό. Για να υπάρξει έγκλημα πολέμου, όπως καταλαβαίνετε πρέπει να υπάρξει πόλεμος. Διεθνής σύραξη μεταξύ κρατών, είτε σύραξης μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ε, ένοπλων δυνάμεων στο εσωτερικό μιας χώρας. Πρόκειται λοιπόν για διαδικασίες οι οποίες ορίζονται επακριβώς αυτό το καταστατικό και φυσικά δεν πρόκειται κάθε φορά για τις ίδιες παραβιάσεις και εγκλήματα. Και στη μία και στην άλλη όμως περίπτωση τα πολιτιστικά αγαθά προστατεύονται γιατί ακριβώς ε, ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία αυτών των αγαθών που προστατεύονται από αυτήν την σύμβαση από τη στιγμή που εντοπίζονται και περιγράφονται σαν πολιτιστικά αγαθά. Θα ξεκινήσω καταρχήν με την πρώτη κατηγορία σειράξεων της διεθνής συγκρούσης για να σας αποδείξω ότι μπορεί σαφώς να διωχθεί αυτή η πράξη και θα αναφερθώ στο άρθρο 8 β9 όπου αναφέρονται εγκλήματα πολέμου ή καθοδήγηση εκ επίθεση κατά μνημείων θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, φιλανθρωπικών, νοσοκομείων, ιστορικών μνημείων και κτηρίων, κτίρια στα οποία συγκεντρώνονται ασθενείς ή τραυματίες. Πρόκειται για επίθεση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Δεν προϋποθέτει αυτό το άρθρο ότι αυτή η επίθεση επιτυχάνει το σκοπό της. Δεύτερον, αυτό το άρθρο διώκει τις επιθέσεις κατά ιστορικών μνημείων. Το καταστατικό της Ρώμης βεβαίως δεν δίνει εδώ ορισμό για το τι είναι ιστορικό μνημείο. Απλώς θα πρέπει το κτίριο του, στο οποίο έγινε η επίθεση να, είναι, ε, να έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα, είτε να ε, βρίσκεται στον κατάλογο των ιστορικών μνημείων της ε, UNESCO. Αυτό είναι μια ένδειξη βεβαίως από τη στιγμή που ένα κτίριο αναγράφεται και περιλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Και αυτή είναι και η προσέγγιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Ιουγκοσλαβία. Επίσης επιθέσεις σε πολιτιστικά μνημεία, κτίρια, όπως παραδείγματο χάρη είναι ένα μουσείο. Τι γίνεται όμως αν η επίθεση στοχεύει τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μνημείου. Βεβαίως εννοείται ότι καταρχήν πρέπει να δούμε την επίθεση στο κτίριο αυτό καθεαυτό, καθότι αυτό αποτελεί το πολιτιστικό κτίριο. Πρόκειται λοιπόν για μια διεθνής, διεθνή προστασία όπως καθορίζεται από τα άρθρα αυτά. Βεβαίως αυτά τα πολιτιστικά αγαθά συμπεριλαμβάνονται στη γενικότερη κατηγορία των προστατευόμενων αγαθών και εδώ αναφέρομαι στις παράγραφους 2, 4, 13 και 16 του άρθρου 8, η παράγραφος 13 αναφέρεται στην καταστροφή, την κατάσχεση τέτοιων αγαθών και διώκει την λαιλασία μιας πόλης είτε ε, μιας τοποθεσίας. Τα πολιτιστικά αγαθά βεβαίως και θα μπορούν να βρίσκονται διασκορπισμένα σε μια τοποθεσία, σε μια πόλη και εδώ διώκεται με μεγάλη σαφήνεια και η λαιλασία αλλά και η κατάσχεσή τους. Σε περίπτωση ε, σειράξεων στο εσωτερικό μιας χώρας, όπως παραδείγματο χάνει το 2012 στο Μαλί, και εδώ προστατεύονται αυτά τα πολιτικά αγαθά σε κάθε περίπτωση όπως ακριβώς και στις διεθνείς συγκρούσεις. Αυτά όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου και στις διεθνείς συγκρούσεις αλλά και στις συγκρούσεις στο εσωτερικό μιας χώρας. Η λαιλασία όμως επίσης προβλέπεται και διώκεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχουν εγκλήματα πολέμου και χωρίς εμπόλεμη σύρεξη. Θα πρέπει όμως να αποδεχτεί ότι υπάρχει συστηματική επίθεση κατά ενός πληθυσμού και καταστροφή πολιτιστικών αγαθών ακριβώς επειδή για πολιτικούς, φιλετικούς, εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς ή άλλους σκοπούς στόχος είναι μια συγκεκριμένη ε, κοινότητα. Όσον αφορά τη γενοκτονία, το καταστατικό της Ρώμης δεν ε, αναφέρει το θέμα της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών σε σχέση με μια γενοκτονία. Όμως η καταστροφή πολιτιστικών αγαθών μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική απόδειξη για το ότι υπάρχει πρόθεση γενοκτονίας. Να επανέλθω τώρα σε λίγο πιο πρακτικά σημεία. Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι χώρες. Υπάρχει καταρχήν η γεωγραφική επικράτεια των κρατών που ανήκουν στο καταστατικό της Ρώμης που έχουν ε, προσυπογράψει 123 χώρες μέχρι τώρα. Στη Συρία και στο Ιράκ παραδείγματο χάρη δεν μπορεί να δράσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γιατί δεν είναι ε, μέλη αυτές οι δύο χώρες. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να έχει αρμοδιότητα εάν αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα ανήκουν σε μια χώρα η οποία έχει προσυπογράψει το καταστατικό της Ρώμης. Δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να δράσει στην Συρία ή στο Ιράκ από τη στιγμή που υπάρχουν στις χώρες αυτές μαχητές που προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γερμανία, μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όσον αφορά την ευθύνη, και εδώ βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η κυρίως υπευθυνη για αυτές τις καταστροφές, στις περιπτώσεις που προανέφερα είναι Ιρακινοί ή Σύριοι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέξει κανείς τους κυρίως υπεύθυνου. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν δραστηριοποιείται σήμερα σε αυτές τις ε, δύο χώρες. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα το Συμβούλιο Ασφαλείας βάσει του κεφαλαίου 7 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών να ε, συλλάβει και να υπάρξει προσαγωγή των υπευθύνων στο ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα πολιτικά αγαθά είναι θέμα και αρμοδιότητα όλων. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που έχετε βάλει το θέμα αυτό στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης. Είναι φυσικά και αρμοδιότητα άλλων φορέων βάσει της αρχής της επικουρικότητας που γνωρίζετε πολύ καλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι όμως και αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η προστασία των πολιτικών αγαθών είναι θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την κυρία Μπενσούντα και την υπηρεσία της. Θεωρούμε ότι το καταστατικό τη Ρώμης προσφέρει δυνατότητε προστασία για την καταπολέμηση αυτή τη μάστιγα, Γνωρίζουμε τι αρμοδιότητε μα σε διεθνέ επίπεδο και έχουμε την πρόθεση να συνεισφέρουμε και εμείς για την καταπολέμηση αυτού του απεχθούς εγκλήματος. Στα πλαίσια αυτά, η υπηρεσία και το γραφείο του Ισαγγελέρ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προετοιμάσει την μεθοδολογία καθώς και τις ε, κοινέ μας δράσεις με όλους τους ε, υπεύθυνους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη νομική βάση, την ισχυρή νομική βάση για αυτήν την ε, δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συνδρομή σας στις εργασίες μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο, να κάνουν ερωτήσεις. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παρουσιάσεις και έχουμε στη διάθεσή μας 20-25 λεπτά για την ε, συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Τρόπελ. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω την ερώτησή μου στον κύριο Λαντζερίνη. Μιλήσατε για την ε, δυνατότητα μιας στρατιωτικής παρέμβασης για να σταματήσει αυτή η καταστροφή πολιτιστικών αγαθών. Μέχρι τώρα όμως δεν υπήρξε πλειοψηφία για να υπάρξει παρέμβαση για διάσωση ανθρώπινων ζώων. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, θα υπάρξει πολιτική πλειοψηφία για την υποστήριξη μιας τέτοιας παρέμβαση για την προστασία των πολιτικών αγαθών. Εάν την ε, φαντάζεστε, τι είδου τέτοια πολιτική ή στρατιωτική παρέμβαση μπορείτε να φανταστείτε επί τόπου για την προστασία των πολιτικών αγαθών. Μπορείτε να μου το περιγράψετε. Κατά την άποψή μου δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και έχω μια ερώτηση για τον ε, κύριο καθηγητή Λαντσερίνη και τον κύριο Καταρχά είπατε ότι χρειάζονται προγράμματα ευαισθητοποίηση για του πολίτε, ε, για του ανθρώπου, έτσι ώστε να ε, έχουν επίγνωση τη αξία τη πολιτισμικής κληρονομία. Και βέβαια το θέμα είναι ότι όταν εγώ μένω σε μια εμπόλεμη κατάσταση, σε μια χώρα όπου γίνεται πόλεμος, είναι βέβαια σημαντικό να προστατεύσω την πολιτισμική μου κληρονομιά, είναι πιο όμως σημαντικό να προστατεύσω τη ζωή μου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το ξέρουμε. Εσείς ποια μέτρα προτείνετε, τι θεωρείτε πως μπορούμε να κάνουμε. Έπειτα προς τον κύριο Τιτέχτχαμ, σχετικά με την συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στο θέμα των ξένων μαχητών. Πώς ε, γίνεται, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έχουμε αρκετές πληροφορίε, έχουμε δει πολλά βίντεο στο διαδίκτυο όπου μέλη της ίσης καταστρέφουν μνημεία σε κληρονομιά. Τι γίνεται, ελέγχεται η κατάσταση, παρακολουθείτε αυτά που συμβαίνουν, μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες από τις εικόνες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ε, γίνονται διώξεις, έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν σε καταστροφή πολιτισμικής κληρονομιάς. Τι ακριβώς συμβαίνει. Κυρία Τζουλί Βόρντ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, πολύ λεπτομερής, γεμάτη πληροφορίες. Αναφερθήκατε σε νομοθεσία, σε πολιτικές, σε τεχνικά ε, μέσα αντιμετώπισης και όλα αυτά τα ακούω σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή διότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο ήμουν στη Σρεμπέντσα όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και να συνομιλήσω με μέλη μιας νέας πρωτοβουλίας της Adopt Σρεμπενίτσα Είναι μια τοπική πρωτοβουλία η οποία προσπαθεί να συγκεντρώσει ε, στοιχεία σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων στην περιοχή αυτή πριν τον πόλεμο. Στην παρουσίασή σας λοιπόν αναφερθήκατε στα κοινοτικά μουσεία, στα μουσεία των, ε, των κοινοτήτων εκεί. όπου φιλοξενούν την ε, πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, την οικογενειακή κληρονομιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναγκάστηκαν να φύγουν ξαφνικά και να, δεν πρόλαβαν καν να πάρουν τα, τις φωτογραφίες τους από το σπίτι, τα ενθύμια της κληρονομιάς αυτής. Αυτά τα ενθύμια δεν έχουν μεγάλη χρηματική αξία, όμως έχουν ανεκτήμητη συναισθηματική αξία για τις κοινότητες αυτές που έχουν χάσει αυτήν την κληρονομιά που υπήρξαν θύματα γενοκτονίας. Όμως η χρηματοδότηση συνήθως πηγαίνει σε πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα και όχι σε αυτά τα ε, μικρά προγράμματα βάσης. Είναι όμως ζωτικής σημασίας η συμβολή τους και η δημιουργία αρχείων τέτοιων και μάλιστα υπό τόσο δύσκολες συνθήκες. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτά τα προγράμματα που είναι τόσο σημαντικά. Έπειτα, αυτές οι πράξεις γενοκτονίας, σε κάποιο σημείο γίνονται και αυτές ε, κομμάτι της ε, πολιτισμικής κληρονομιάς, μιας δύσκολης πολιτισμικής κληρονομιάς. Εμείς πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτό το μέρος της ε, πολιτισμικής κληρονομιάς, διότι κάποιοι προσπαθούν να καταστρέψουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία όμως αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής αυτής αποτελούν ε, και εκείνα πολιτισμική κληρονομιά. Χρειάζεται να το συζητήσουμε, διότι πολλές φορές αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες έτσι ώστε να μάθουν οι επόμενες γενιές το τι συνέβη και να αποτρέψουν να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Η Οστρογεύκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτή της ε, συζήτησης. Ήμουν ε, από αυτού που ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί, καταρχήν, γιατί θα ήθελα να διαπιστώσουμε το μέγεθος αυτού του φαινομένου. Και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση. Σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η ψηφιακή κατάταξη και αρχαιοθέτηση αυτών των πολιτιστικών αγαθών που είτε καταστράφηκαν είτε καταστρέφονται και θα πρέπει σίγουρα να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες αυτής της κατάταξης σε ψηφιακά αρχεία. Είτε πρόκειται για καταστροφές εκ προθέσεως, είτε πρόκειται για καταστροφές οι οποίες συνεχίζουν να συμβαίνουν από αμέλεια. Είναι αλήθεια ότι σήμερα στην Αφρική παιδιά πεθαίνουν από έλλειψη νερού. Ολόκληρα χωριά εξαφανίζονται από το χάρτη, καταστρέφονται και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ευαισθητοποιήσει κανείς την κοινή γνώμη και να στηρίξει δράσεις για την προστασία των ε, πολιτιστικών αγαθών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε ε, πληθυσμούς. Επίσης, όσον αφορά τα γεγονότα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, θυμόμαστε όλοι αυτά που συνέβησαν εκεί και γι' αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ την καταστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποια μνημεία καταστρέφονται γιατί θεωρούνται σαν ε, στρατιωτικός στόχος. Παραδείγματος χάρη πρέπει να καταστραφεί μία γέφυρα για να εμποδιστεί η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τη Συρία όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται για στρατιωτικούς στόχους, πρόκειται για λαιλασία, για καταστροφή, η οποία είναι αυτός σκοπός για να καταστραφεί η πολιτιστική κληρονομιά μιας κοινωνίας, κάτι που είναι καθοριστικό οι εμπειρογνώμονες εξάλλου έχουν υπογραμμίσει αυτό το χαρακτηριστικό αυτών των καταστροφών και θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω ποιος είναι ο προϋπολογισμός ε, του ΙΡΚΟΜ. Και μία άλλη ερώτηση. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ποιοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Διαθέτουμε ψηφιακά αρχεία και φωτογραφίες όλων αυτών των μνημείων που καταστράφηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι σήμερα συζητούμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και να σας ευχαριστήσω επίσης για τους προσκεκλημένους οι οποίοι μας ε, παρουσίασαν την ε, δική τους άποψη σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Με χαρά μου παρατήρησα ότι έχει δημιουργηθεί μία ε, μονάδα στην Χάγη για το συγκεκριμένο θέμα με επιτυχία. Όμως πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους ορισμούς. όχι μόνο με τον ορισμό της πολιτισμικής γενοκτονίας, αλλά και με την ίδια τη γενοκτονία. Οι ορισμοί δεν είναι σαφείς και είναι διαβλητοί. Πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε τον ορισμό της γενοκτονίας σε όλα τα γεγονότα όπου για πολιτικούς λόγους έχουν σημειωθεί για παράδειγμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945. Ε, έχουμε συζητήσει αρκετά για την Σρεμπρένιτσα, όμως πρέπει να μην ξεχνάμε και όσους έχασαν τη ζωή τους στην πρώην Γεκοσλαβία όταν οι κομμουνιστικές δυνάμεις ανέλαβαν την ηγεσία στην περιοχή. Και δεν πρόκειται μόνο για ένα έθνος, αλλά 7-8 διαφορετικά έθνη τα οποία προήλθαν από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Σύμφωνα λοιπόν με τον υφιστάμενο ορισμό, αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν περιπτώσεις γενοκτονίας. Τόσο το καταστατικό της Ρώμης όσο και τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζεται να επεκτείνουν τον ορισμό της γενοκτονίας και πρέπει επίσης να συζητήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της καταστροφής της πολιτισμικής κληρονομιάς. Δεν είναι απαραίτητα έγκλημα πολέμου, όμως χρειάζεται να το συζητήσουμε. Η κυρία Μπίλτ. Σας ευχαριστώ. Για την Παλμύρα στη Συρία έχω μια ερώτηση και είχαμε υποβάλει και μια πρόταση ψηφίσματος ζητώντας ε, την προστασία αυτού του μνημείου, αυτής, αυτού του στοιχείου πολιτικής κληρονομιάς. Δεν ξέρω λοιπόν σε ποιο βαθμό έχουμε έρθει σε επαφή, σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Συρία προκειμένου να προστατεύσουμε ακριβώς αυτά τα κοιμήλια προστατικής ε, κληρονομιάς. Ε, ο κύριος Μόργανο, ευχαριστώ πρόεδρε. Να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου. Καταρχάς για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής, τις παρουσιάσεις που είχαμε σήμερα, τις συνεισφορές, οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα ε, τόνισαν μια σειρά από πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι επί της ε, πολιτικής επιλογής και βουλήσεως η εστίαση, η συγκεκριμένη στα πράγματα, η έρευνα θα έλεγε κανείς με το μικροσκόπιο για να ε, έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία και λεπτομέρειες για κάθε ένα από αυτά τα εγκλήματα της πράξης αυτές είναι απόλυτα χρήσιμη. Αλλά έχω μια διτή ερώτηση επί δύο πτυχών. Καταρχάς έχουμε την ε, προληπτική δράση. Έχουμε μια ολόκληρη προσπάθεια κατάρτισης και εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης αν θέλετε. Δηλαδή αυτοί που αυτή τη στιγμή ζουν δίπλα σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να αντιλαμβάνονται την αξία των στοιχείων αυτών. Και αυτό είναι μια προσπάθεια που θα πρέπει να είναι όλο και πιο στοχευμένη. Γιατί πρόκειται για μια βοήθεια να κατανοήσει κανείς την αξία ενός ε, στοιχείου, ενός κοιμηλίου, ενός αγαθού που είναι σημαντικό για το σύνολο της ανθρωπότητας. Εγώ όμως προσπαθώ να καταλάβω λίγο καλύτερα, καθότι έχουμε και μια νομική εστίαση, γιατί αυτές οι πράξεις, ε, πέρα από καταστροφή και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο σήμερα. Γιατί πέρα από την καταστροφή έχουμε και το παράνομο εμπόριο και τη διάθεση την παράνομη αυτών των κοιμηλίων, αυτών των αγαθών, αυτών των στοιχείων. Και γνωρίζουμε ποιε είναι οι αγορές εντός αγωγικών που δραστηριοποιούνται σε αυτό και αγοράζουν. Εκεί έρχεται και η δική μας δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση και επομένως το νομοθετικό πλαίσιο που να πηγαίνει πολύ πέρα των εθνικών συνόρων, ορίων νομικών, γιατί έχουμε κλοπή, και έχουμε παράνομη διάθεση και τελικά παράνομη αγορά εκείνων που τελικά αποκτούν με τον παράνομο τρόπο αυτά τα στοιχεία. Λέγω αυτό διότι οι συνάδελφοι υπογράμμισαν όλα τα υπόλοιπα θετικά στοιχεία και καλά έκαναν, αλλά ίσως αυτή εδώ η πτυχή θα πρέπει να φωτιστεί λίγο περισσότερο και να διαρευνηθεί λίγο περισσότερο. Και ίσως δεδομένης και της επικαιρότητα των εξελίξεων θα πρέπει να καλύψουμε το κενό αυτό για να μπορέσουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ. Με αυτό το τελευταίο ερώτημα λέει ο Πρόεδρος. Δίνω αμέσως το λόγο για τις απαντήσεις ε, στα μέλη του πάνελ. Ήθελα και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση. Και προς τους δύο καθηγητές. Η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα θα ήθελα να καταλάβω πώς έχει ενεργοποιηθεί γιατί μιλούμε για την ε, Ίκραμ, ε, Ίκρομ, με και μια τεχνική αν θέλετε δραστηριοποίηση, αλλά εδώ θα μπορούσαμε να μπούμε και σε ύδατα συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημιακών φορέων. Υπάρχει ένα δίκτυο της Μεσογείου, για παράδειγμα ακαδημαϊκό. Επομένως και σε αυτό το επίπεδο για έναν καλύτερο συντονισμό για τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης πέρα από τα έγγραφα δηλαδή που παράγονται. Ήθελα να καταλάβω κατά πόσον υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της ΣΥΚΡΟΜ και των πανεπιστημιακών φορέων. Το άλλο που ήθελα να υπογραμμίσω είναι το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι και συμφωνώ. Από τη στιγμή κατά την οποία μπορεί να πει κανεί ότι έχουμε τις νομικές βάσεις, το νομικό πλαίσιο, εσείς ε, κύριε Ντουτέχτχο θεωρείτε ότι Έχουμε μια ανάγκη νέου, ορισμού της αρμοδιότητας του δικαστηρίο, μήπως. Διότι και οι νομικές συνέπειες όλων αυτών των δράσεων ή των εγκληματικών δράσεων Ας ακούσουμε με τη σειρά πρώτα τον κύριο Λεντζερίνη, αν θέλετε, και μετά τους υπόλοιπους, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε σε 10 λεπτά, το κατα, κατά μέγιστο μου λένε. Δεν έχουμε πάνω από 10 λεπτά. Γιατί έχουμε και το δεύτερο πάνελ λοιπόν, και να μην τους κλέψουμε το χρόνο. Για τη λαθρεμπορία, αν δεν σας πειράζει, να αφήσουμε το λόγο στο επόμενο πάνελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις σε λίγα λεπτά. Το θέμα της πολεμικής ε, παρέμβασης υπήρξε αντιφατικό εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου και της χρήσης ε, της βίας των όπλων για την επίλυση διεθνών προβλημάτων. Βεβαίως η πολεμική παρέμβαση σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από την προστασία των ανθρώπων. Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη. Σήμερα μιλούμε για την πολιτική κληρονομιά και έτσι εστιάστηκα και εγώ σε αυτό αλλά είναι σαφές ότι όλα τα εγκλήματα που διαπράττει η ISIS και άλλες ομάδες είναι διασυνδεδεμένα. Και με τον κύριο Ντεκάρο μιλούσαμε για αυτήν την υποκειμενική έννοια, αν θέλετε, η αντίληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς που πηγαίνει πολύ πέραν της συμβάσεως της διεθνούς πολιτικής κληρονομιάς σχετικά με τα μνημεία εξαιρετική αξία κτλ. κτλ. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η αντίληψη των μεμονωμένων κοινοτήτων και ομάδων για την δική τους πολιτιστική κληρονομιά και γι' αυτό μιλούμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι καταστρέφουν τα κοιμήλια της κληρονομιάς. Την ίδια την ταυτότητα την πολιτιστική και πολιτισμική θέλουν να καταστρέψουν. Και επομένως αυτά που είναι σύμβολα μιας άλλης ομάδας, μιας άλλης κοινότητας. Άρα με οποιαδήποτε παρέμβαση προστατεύει κανείς την ε, πολιτιστική κληρονομιά ως βασικό στοιχείο ταυτότητας και ταυτόχρονα την υλική ταυτότητα, τα υλικά σύμβολα της επιβίωσης της σωματικής πλέον των ομάδων αυτών. Και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι όλες αυτές οι δράσεις γίνονται σκοπίμως με πρόθεση να οδηγήσουν σε μια κλιμάκωση τι είδος πολεμικής παρέμβασης. Αυτό μπορεί να το συζητήσει κανείς. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα παρέμβασης. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει η πολιτική βούληση, η πολιτική θέληση και πρέπει να διοργανώνεται οποιαδήποτε παρέμβαση και να διεξάγεται προς τις συνθήκες, ανάλογα με τις συνθήκες του συγκεκριμένου κρούσματος επεισοδίου και σε συνεργασία με αυτούς που μάχονται για να υπερασπιστούν το έδαφος τους, την κοινότητά τους ή το σύμβολο της ταυτότητός τους. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, στι διεθνείς διαπραγματεύσεις να χρησιμοποιούμε, να θα περισσότερο με, τους, με τις ομάδες των Κούρδων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι οι μόνοι που μάχονται με το όπλο στο χέρι κατά της ISIS. Θα μπορούσε λοιπόν μια, ένα πρώτο επίπεδο παρέμβασης να αφορά σε τέτοιες δράσεις στήριξης. Τώρα για τον ορισμό της γενοκτονίας συμφωνώ ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τον ορισμό αυτόν για να συμπεριλάβουμε και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ακριβώς όπως είναι και η πρόθεση των δραστών. Και νομικώς μιλώντας, έχουμε μια σύμβαση επί της γενοκτονίας, έχει υιοθετηθεί από το 48 και σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, τη συνθήκη αυτή, η γενοκτονία είναι μόνο η φυσική καταστροφή της κοινότητας το διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο που είναι η πιο σημαντική διεθνή αρχή στην ερμηνεία του διεθνούς δικαίου επαναλαμβάνει ότι εκεί περιορίζει την ερμηνεία της ή στη φυσική, σωματική αν θέλετε καταστροφή ενώ όταν έχουμε ακριβώς αυτό μάλλον εννοούσα όταν έλεγα ότι η καταστροφή της πολιτιστική κληρονομιάς είναι ένδειξη τέτοια προθέσεω, και αυτό νομίζω θεωρούσε και το δικαστήριο δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο η πιο προκεχωρημένη θέση πρέπει να συμπεριλαμβάνει την καταστροφή της πολιτικής κληρονομιάς και ταυτότητας, θεωρώ, σε προσωπικό επίπεδο όμως. Νομικά είναι λίγο πιο περίπλοκο να το στοιχειοθετήσει κανείς αυτό. Για την ε, ευαισθητοποίηση, ο κύριος Ντεκάρο αναφέρθηκε στην ευαισθητοποίηση των, ε, του πληθυσμού των ομάδων για την αξία της παραδοσής τους και της ε, ηλικής τους και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και είναι προφανές ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς περισσότερο ενδιαφέρονται να βρουν τροφή παρά να προστατεύσουν την ταυτότητά τους. Αλλά ευαισθητοποίηση σημαίνει να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι ακριβώς η πολιτιστική κληρονομιά είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ε, υπόστασής τους και της ηλική. διότι διαφορετικά θα καταστραφεί αυτή η έννοια και για αυτούς και για τις μελλοντικές γενναίες. Σας παρακαλώ να είστε λίγο συντομότεροι γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Τικάρο. Μία συλλογική απάντηση πιθανώς και συνοπτική γιατί είναι αδύνατο να απαντήσω στα πάντα. Είμαστε υπό την επίρρεια τρόπον δεινά της ε, συμβάσεως UNESCO του 1972, η οποία καθυστέρησε να έρθει στην ιστορία της UNESCO. Η έννοια της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς πηγαίνει πολύ πέραν του καταλόγου των στοιχείων της πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς, οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν ως σημαίες, αν θέλετε, σύμβολα των βελτίστων πρακτικών του συνόλου. Τώρα, η πολιτική υπογράμμιση που έχει δοθεί στις συγκεκριμένες, στα συγκεκριμένα πεδία πολιτιστικής κληρονομιάς σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τονίζουμε την Παλμύρα και όχι τα υπόλοιπα 50 σημεία τα γεωγραφικά που έχουν πληγεί. Όμως αν δείτε την εγγραφή ή στον κατάλογο αυτών, αυτή έχει οδηγήσει σε στόχευση, σε μια λίστα στόχων. Γιατί αν θέλω να δηλώσω την πολεμική μου ικανότητα, θα πλήξω το στόχο εκείνο που συμπεριλαμβάνεται σε ένα κατάλογο. Και επομένως από την έννοια αυτή έχει επικοινωνιακή μεγάλη σημασία ο κατάλογος αυτός. Όμως η ίδια η κληρονομιά που βασίζεται στο, σε μια συλλογική μνήμη και εκπαιδευτικό επίπεδο είναι κάτι πολύ πιο ασαφές και ευρύ και άειλο. Υπό την έννοια λοιπόν της χρήσης ε, της επικοινωνιακής τακτικής και των ε, λεγόμενων universal values, όπως και το, το ανεπίλητο θέμα της εθνικής ταυτότητος όλες τις χώρες μας, στην Ιταλία, στη Γερμανία, όπου θέλετε, προερχόμαστε από τάσεις του 1800 και 1900 που οδήγησε στην ιδέα του έθνους κατά πλήττοντας, καταστρέφοντας την πιο συλλογική ιδέα της συλλογικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς και αγαθού και αξίας. Το, θέτοντας τη μία ιδέα πολιτιστικής κληρονομιάς κατά της άλλης. Ενώ η ιδέα της UNESCO είναι sharing in diversity. Δηλαδή το πώς μπορούμε να μοιραστούμε τις διαφορετικές αυτές ιδέες και έννοιες. Και όχι να πούμε ότι η χ ταυτότητα αντιπαρατίθεται προς την ψ. Βεβαίως και έχουμε πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά το να χρησιμοποιούμε τα κίνητρα ή τις αιτίες ενός πολέμου για να υπερασπιστούμε μια εθνική ταυτότητα είναι να οδηγούμε στον επόμενο πόλεμο. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι κάτι αρκετά περίπλοκο και πολυεπίπεδο που συμπεριλαμβάνει διάφορες ταυτότητες. Για τέλος, ποιος θα υπερασπιστεί το Κολοσσέο. Οι Κινέζοι που είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ε, ε απέναντί μας έχουμε ένα μέλλον πολύ πιο περίπλοκο από εκείνο του 19ου αιώνα, από τις ιδέες του ρωματισμού, της εθνικότητας του εθνικισμού. Πρέπει η παγκοσμιότητα να γίνει αντιληπτό ότι είναι μια έννοια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντουτέχτρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν. Η προστασία από τους ίδιους τους πληθυσμούς των πολιτιστικών αγαθών, ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι απειλούνται, απειλεί τη ζωή τους. Και θα πάρω σαν παράδειγμα το μαλλί. Δεν είναι τίποτα εμπιστευτικό αυτό που θα πω, είναι γνωστά τα στοιχεία οι κάτοικοι αυτής της περιοχής ε, εν μέσω ένοπλων σειράξεων προστάτευσαν κάποια χειρόγραφα και βιβλία που βρισκόταν σε συγκεκριμένους χώρους και βιβλιοθήκες. Και σε πολλές δύσκολες λοιπόν περιοχές όπως του Μπουκτού ενώ υπήρχε ε, κατοχή αυτό συνεχίστηκε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και όλοι ξέρουμε ότι τα στοιχεία που διαθέτει το ποινικό δικαστήριο σήμερα μας επιτρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, τι κάνει το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παρακολουθήσει όλους αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν να φύγουν από την Ευρώπη, παραδείγματο χάνει, για να πάνε ε, να πολεμήσουν στη Συρία. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή ε, εντοπισμός από τα κράτη Βεβαίως υπάρχουν σήμερα πολλά μέσα στη διαθεσή μας για να εντοπίσουμε τα άτομα αυτά, τα οχήματα που χρησιμοποιούν και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό όμως είναι θέμα τεχνολογίας. Μιλήσατε και για το θέμα της ε, ψηφιακής αρχαιοθέτησης. Επίσης μπορούμε σήμερα να έχουμε τρισδιάστατες απεικονίσεις αυτών των μνημείων που έχουν καταστραφεί και να δείξουμε τις, ε, επόμενες γενιές παραδείγματο χάρη πώς ήταν αυτό το μνημείο και να αποδείξουμε εν ότι καταστράφηκε ή ότι καταστράφηκε εν μέρη. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα κάτι που μπορεί να μπει στην κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου. Είναι πολύ σημαντικό όμως γιατί σήμερα διαθέτουμε αυτά τα λογισμικά και μπορούμε βάσει στοιχείων να απεικονίσουμε τα μνημεία αυτά εάν έχουν κατασταθεί. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε επίσης και για το θέμα της γενοκτονίας. Τι διαθέτουμε σήμερα, τι διαθέτει το Διεθνές Ποινικό Δικαστηρίο για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επιθέσεων και λαιλασίας αλλά και κατάσχεσης πολιτικών αγαθών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα δίεξη αυτών των προσώπων. Ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα για την περίπτωση των γεγονότων στο Μάλι και φυσικά εδώ αυτό γίνεται με την συμμετοχή των κρατών. Φυσικά και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη πρέπει το θέμα της γενοκτονίας να μπορέσει να συνδεθεί με την καταστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Γιατί ουσιαστικά καταστρέφονται κάποια στοιχεία της ιστορίας και της ε, κληρονομιάς της πολιτιστικής έτσι ώστε να μην μπορέσουν οι επόμενες γενιές να αναγνωρίσουν την ιστορία τους και την ταυτότητά τους. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει μια μεταρρύθμιση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να συμπεριληφθεί και αυτό το έγκλημα. Ευχαριστώ όλους ε, τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Εκτός από τις συνεισφορές σας έχουμε και τις ε, γραπτές παρουσιάσεις, θα τις ε, και αν θέλετε να καθίσετε στα έδρανα της ΕΦΣΑ για να προσκαλέσω τους επόμενους, την επόμενη ομάδα και για να κερδίσουμε χρόνο καθότι έχουν καθυστερήσει λίγο να σας τους παρουσιάσω. Παρακαλώ. Okay. Allora, eh, Λοιπόν, το δεύτερο πάνελ, όπως γνωρίζετε, είναι αφιερωμένο στο λαθρεμπόριο αγαθών πολιτιστικής ε, κλονιάς. Είχαμε δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ασφαλείας ε, του 2013 και του 2015, ένα που αφορούσε στη Συρία και άλλο στο Ιράκ και στα οποία προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, τι κενά έχουμε, τι ελλείψεις. Allora, noi abbiamo Λοιπόν, να παρουσιάσω λοιπόν συμμετέχοντας ο κύριος Μάρκ Αντρέ Γονού από το Κέντρο Τεχνών και Δικαίου του Μονεστήνου της Γενέβης σχετικά με την παράνομη διάθεση των αγαθών πολιτικής οικονομίας και ο κύριος Εντουαρ Πλόνς της UNESCO και ο κύριος Φαμπρίτσιο Πανόνε της Ίντερπολ και με αυτή τη σειρά παρακαλώ να έχουμε τις παρουσιάσεις. Παρακαλώ τον κύριο Γονό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Εδώ συνοψίζουμε με την παρουσίαση αυτή πολλά από τα θέματα ε, που ήδη θίξαμε, των συγκρούσεων, των σειράξεων, των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε στη Συρία και στο Ιράκ. Καταρχά να τα δει κανεί ε, στο πλαίσιο του τι μπορούμε να κάνουμε εδώ ω Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπω τρία σημεία, τρία μέτρα. Μέτρα στο πεδίο, μέτρα για την εισαγωγή και μέτρα για την αποκατάσταση ή επιστροφή των στοιχείων αυτών. Συνοψίζω σε δύο λόγια το υπάρχον νομικό πλαίσιο που βασίζεται σε συμβάσεις που ήδη ακούσαμε. Ο κύριος ε, Πλόνς θα σας πει περισσότερα. Έχουμε την σύμβαση του 70, του 95 και άλλα σημαντικά κείμενα της Χάγης του 54 και ένα πολύ πρόσφατο πρωτόκολλο που αφορά στην ε, πρόληψη του, της λαθρεμπορίας κατόπιν κα, ε, κατοχής, δηλαδή κατεχομένων ζωνών. Και μετά είχαμε και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, ε, του 99. Δηλαδή έχουμε μια, ένα, μια ευρεία δέσμη νομικών μέσων στη διαθέσή μας. Τώρα πιο συγκεκριμένα. Για τα μέτρα μπορούν να ληφθούν επιτόπου πρέπει να διευκολύνουμε την εφαρμογή του ούτω ώστε να προλαμβάνουμε όλα αυτά τα κρούσματα λαθρεμπορίας. Τι μπορεί να κάνει η Αραγική Ένωση? Να συνεργαστεί στην επιτήρηση και φύλαξη των μουσείων και μνημείων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους ε, κρίσεως, απειλής δηλαδή, κατά των μνημείων αυτών. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές το παράδειγμα, αλλά στο Μαλή η κοινωνία των πολιτών συμμετείχε ενεργά στην προστασία κοιμηλίων, χειρογράφων από το Τιμπουκτού, για παράδειγμα. Όταν λοιπόν η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει ενεργά, μπορεί να επιτύχει πολλά. Επίσης μπορούμε να φανταστούμε την εφαρμογή αυτών που ονομάζουμε στα αγγλικά ασφαλείς λιμένες safe havens, όπου ή στο πεδίο και στο εξωτερικό μπορούν να υλοποιηθούν για να προστατεύσουν τα κοιμήλια αυτά. Και πρόσφατος, ε, και ζητώ συγγνώμη ε, ως Ελβετός ε, εκπρόσωπος εδώ, αλλά στην Ελβετία γράφει στην Εθνική Νομοθεσία ότι η προστασία των κοιμηλίων κατόπιν καταστροφής, πολεμικών σειράξεων κτλ. επιτρέπει τη δημιουργία safe haven ασφαλών λοιπόν λιμένων ή αν θέλετε χώρων φύλαξης αυτών των αγαθών των κοιμηλίων. Δεύτερον, ο έλεγχος στα σημεία εισαγωγή. Ένας αυστηρός έλεγχος ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε αυτή τη στιγμή έναν έλεγχο εξαγωγικό υιοθετήθηκε κανονισμός που επιτρέπει τους εξαγωγικούς ελέγχους αλλά για τους εισαγωγικούς ελέγχους δεν έχουμε και πολλά πράγματα για θέση μα. Και ε, θα λέει κανείς, ε, πρώτη ανάγνωση, κανονικό είναι. Θέλουμε να ελέγξουμε αυτά που βγαίνουν παρά αυτά που μπαίνουν. Αλλά για τι ζώνες κινδύνου όπως είναι το Ιράκ και η Συρία αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι είναι θεμελιώδη σημασία να εφαρμοστούν τέτοιε διατάξει, τέτοια μέσα. Και είναι ένα από τα αντικείμενα του ψηφίσματό σα, δηλαδή να υλοποιηθούν τέτοιοι έλεγχοι. Και δεν είναι και τόσο περίπλοκοι ε, στην εφαρμογή τους. Θα πρέπει οι Ιταλονιακές και οι αστυνομικές αρχές να απαιτούν την παρουσία που θα συνοδεύει το αγαθό ενός πιστοποιητικού και αν δεν υφίσταται δεν θα μπορεί να εισαχθεί. Δηλαδή θα υπάρχει μια προϋπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας. Βεβαίω έχουμε διμερεί συγκεκριμένε σχέσει μεταξύ κάποιων χωρών, όπου συμπεριλαμβάνονται τέτοιε διατάξει, αλλά αυτό θα μπορούσε να γενικευθεί για να καλύπτει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι χωρών όπω ακριβώ η Συρία και το Ιράκ. Και τρίτον, στην περίπτωση μια παράνομη εισαγωγή, εφόσον δεν μπορέσαμε να την παρεμποδίσουμε, θα πρέπει να προβλέπουμε ένα σύστημα αποκατάστασης, επιστροφής δηλαδή, προς τη χώρα προέλευσης. Σύμφωνα με τα όσα ε, προβλέψατε στο ευρωπαϊκό σας δίκαιο, μέσω της οδηγίας επιστροφής που προσφάτως επανεξετάστηκε αναθεωρήθηκε. Στο άρθρο 5 υπό τη σύμβαση του 95. Δηλαδή, τι θα κάναμε εκεί. Θα δημιουργούσαμε, θα προετοιμάζαμε, θα ολοκληρώναμε ένα σύστημα που θα προέλευε την επιστροφή του αγαθού στη χώρα προέλευσής τους, ας πούμε τη Συρία ή το Ιράκ, επί παραδείγματι, πρόκειται για ένα αρχαιολογικό έβριμα ή είναι άλλο αγαθό υψηλής πολιτιστικής αξίας και αυτομάτως θα ειδίδεται η νομική δυνατότητα της επιστροφής. Και νομίζω ότι αυτέ οι διατάξει που τι έχουμε στα πλαίσια συγκεκριμένων συμφωνιών θα έπρεπε να τι διευρύνουμε. Τώρα πρέπει να το κάνουμε αμέσω, ή πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα σειράξεων. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να φανταστεί κανεί εύκολα ένα σύστημα ασφαλού φύλαξη, safe haven τέλο πάντων, προτού επιστραφούν στον νόμιμο κατοχό του αν θέλετε να το πούμε έτσι. και χώρες που έχουν υιοθετήσει τέτοια στήματα είδαν, είδαν την εμφάνιση περιπτώσεων εθελοντικής επιστροφής τέτοιων αντικειμένων. Διότι αυτοί που τα κατέχουν παρανόμως, με το φόβο των κυρώσεων που προβλέπει το σύστημα, τελικά σε πολλές περιπτώσεις τα επιτρέφουν εθελοντικά. Στη Γενέβη είχαμε μία περίπτωση ενός αναγλήφου το οποίο επιστράφει από είχε κλαπεί από την Νίμρουντ και, και επιστράφει υπό το φόβο των ε, σοβαρότατων κυρώσεων που θα είχε σε περίπτωση που παρέμενε στην παράνομη κατοχή του. Αν λοιπόν, αν λοιπόν συνεργαστούμε στην ε, ασφαλή φύλαξη, στους ασφαλείς λιμένες, στα, ε, στους εισαγωγικούς ελέγχους και προδέσουμε επιστροφές, θα έχουμε ήδη υλοποιήσει πάρα πολλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ και για τη σαφήνειά σα και για την και για τις προτάσεις σας τις πολύ συγκεκριμένε. Ο κύριος Εντουάρ Πλάνς που εκπροσωπεί την UNESCO για την παρακολούθηση της συμβάσεως ε, της UNESCO ακριβώς του 70 για τα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ακριβώς της ε, λαθρεμπορίας και της λαθρέας εισαγωγής στοιχείων κληρονομιάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ήδη είχατε καλέσει την UNESCO σαν ε, εταίρσος για την προετοιμασία και τις ακροάσεις ε, για την σύσταση της οδηγίας. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή για τα όσα έκανε είναι κάτι που πραγματικά μας δίνει δύναμη. Θα ήθελα εξ ονόματος της Γενικής Διευθύντριας κυρίας Μπόκοβα της UNESCO να στηρίξω όλες σας τις προσπάθειες και την ίδια ώρα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα σύνολο κανόνων έξι συμβάσεις επί των οποίων στηρίζεται η δράση της UNESCO για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών το 1995. Υπάρχει η σύμβαση αυτή. Σήμερα η σύμβαση αυτή του 70 που είναι η, νομική, η βασική νομική βάση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών μετέχουν 129 χώρες. Η τελευταία είναι το Λουξεμβούργο που προσχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ιρλανδία, η Λετωνία και η Μάλτα είναι τρει χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα δεν έχουν προσχωρήσει. Ελπίζουμε μέχρι το τέλο του χρόνου αυτό να συμβεί. Και έτσι θα είναι εξαιρετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού όλα τα μέλη της θα έχουν προσυπογράψει. Βλέπετε εδώ ποιοι είναι αυτοί που έχουν κυρώσει αυτήν την σύμβαση. Πρόκειται κυρίως για χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτά τα αγαθά και όχι οι χώρες διακίνησης. Διαπιστώνεται επίσης ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό για την ανάκτηση και την επιστροφή αυτών των αγαθών. Σήμερα συνεχίζουν τα φαινόμενα λαιλασίας και τα τάσχεσης αυτών των αγαθών, οι εμπόλεμες σειράξεις. Περιμένουμε τα κράτη το ταχύτερο δυνατόν, όσοι δεν το έχουν κάνει, να ακυρώσουν αυτή τη σύμβαση, διότι επαναλαμβάνω αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η προσπάθεια, ιδιαίτερα μέσω του δικτύου KILT.net και μέσω του μηχανισμού JAES, μηχανισμό στήριξης. Πέρσι στο Μαρακές και με συμμετοχή αφρικανικών χωρών για την παράνομη διακίνηση τέτοιων πολιτικών αγαθών στην Αφρική. Συναντηθήκαμε για την προστασία επίσης ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία, ένα πρόγραμμα με σημαντικά ποσά, 2 εκατομμύρια ευρώ παραδείγματος χάρη για το 2014 με σκοπό βεβαίως ε, την ειρήνευση της περιοχής και την προστασία των πολιτικών αγαθών καθόν και την βιώσιμη ανάπτυξη της ε, χώρας αυτής. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο βεβαίως καθοδηγείται από τη Βηρητό με συνεργασία και άλλων εταίρων, το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο που συνεισφέρει και μας επιτρέπει να έχουμε άμεση άποψη για το τι γίνεται επί τόπου, λαϊλασίες, καταστροφές και για τα μνημεία που εγγράφονται στην πολιτική κληρονομιά την παγκόσμια, αλλά και σε βεβαίω αρχαιολογικούς χώρους που ξέρετε ότι είναι στόχοι αυτών των καταστροφών, αλλά και βεβαίως της άλλη πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ πρόσφατες ε, δράσεις της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καταστροφή που λαμβάνει η χώρα στην Παλμύρα όπως ξέρετε αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται με την καταστροφή μνημείων και συγκεκριμένων κτηρίων τεμέν τα οποία έχουν καταστραφεί στην περιοχή και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε όλους αυτούς που προστατεύουν επιτόπου την πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή αυτή της Συρίας μεταφέροντας ε, έργα τέχνης από τα μουσεία παρόλο που υπήρξαν και κάποιες καταστροφές και μέσα στα μουσεία. Αυτή η εταιρική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ UNESCO και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται, όπως ξέρετε, μέσω εμπειρογνωμόνων το περίφημο ρόστερ με 120 εμπειρογνώμονες πρόκειται για ένα ασφαλές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών. Μπορείτε όλοι να κάνετε αίτηση στο διαδίκτυο και να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο αυτό. Το παρατηρητήριο, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είναι καθόλου ευανάγνωστα αυτά που σας παρουσιάζω στις διαφάνειες, Έχουμε λοιπόν το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων δίκτυα ασφαλή ανταλλαγής πληροφοριών και βεβαίως πολύ συγκεκριμένες συναντήσεις και workshop ε, για την ε, προστασία των πολιτιστικών αγαθών τον Οκτώβριο του 2014 στο Χαλέπι, προστασία των μουσείων, βάση δεδομένων για τα κλεμμένα έργα τέχνης, ενημέρωση για τις ε, τελωνιακές αρχές ε, και για τις ε, διασυνοριακές δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ αρχών των κρατών μελών. Όπως ξέρετε η διακίνηση αφορά πολλά κράτη και βεβαίως το θέμα της προστασίας της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορείτε να δείτε εδώ αυτά τα σεμινάρια κατάρτισης. Πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν στη Συρία και στις γειτονικές χώρες. Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO έχει κινητοποιήσει όλους τους εταίρους. Ιντερπολ βεβαίως, Διεθνής Οργάνωση Τελωνίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συμμετοχή βεβαίως και κινητοποίηση των ε, τελωνιακών αρχών και βεβαίως την UNEDIC και άλλους φορείς και οργανισμούς των Ηνωμένων Αθηνών, ΙΚΡΟΜ, ΙΚΟΣΜΟΣ, βάσει του ψηφίσματος 2199, κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία και προσπάθεια για την προστασία των αγαθών πολιτιστικών αγαθών συγγνώμη, και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γνωρίζετε την έκθεση που έχουμε προετοιμάσει και φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί με πολύ συγκεκριμένες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται συχνά στην οδηγία καθώς και στις δράσεις που έχουν αναλυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρωματικά με την εθνική πολιτική των κρατών μελών. Ολοκληρώνω αναφερόμενος στις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε. Καταρχήν ε, διάδοση πληροφοριών. Αυτές που περνούν ε, στα δίκτυα της UNESCO μέσω της Interpol, παραδείγματο χάρη, Ξέρουμε ότι παραδείγματο χάρη κάποια αντικείμενα έχουν κλαπεί, δεν ξέρουμε όμως πώς διακινήθηκαν, πού πάνε. Και βεβαίως τα μνημεία αναφέρουν την απώλεια κάποιων ε, αντικειμένων. Υπάρχει όμως μια πολύ συγκεκριμένη διάθεση στη μαύρη αγορά, στις ιδιωτικές συλλογέ και όλοι αυτοί οι οποίοι πολλούν και αγοράζουν παράνομα αυτά τα έργα τέχνης. Πολλές φορές ε, αυτά τα αντικείμενα τα ξαναβρίσκουμε 10-20 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά πλαστά αντίγραφα έργων τέχνης. Ξέρετε ότι αυτό το εμπόριο σαφώς και χρηματοδοτεί τους τρομοκράτες αλλά και κάποιους άλλους έμπορους τέχνης σε κάθε περίπτωση η πολιτική μας θα πρέπει να ενισχυθεί με καλύτερη συνεργασία, με την απαγόρευση αυτών των εξαγωγών. Επαναλαμβάνω υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα και πλαστά αντικείμενα στην αγορά αυτή. Και αναφερόμαστε σε χιλιάδες μικρά αντικείμενα τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να διακινηθούν, να πολιθούν μέσω των ε, ιστοσελίδων λαθρεμπορίου έργων τέχνης. Ενίσχυση λοιπόν των εθνικών νομοθεσιών, των ποινικών, της ποινική δίωξης και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια της σύμβασης της Χάγης και του δεύτερου πρωτόκολλου, το οποίο δεν έχει ακόμα δυστυχώς κυρωθεί από αρκετά κράτη-μέλη και εδώ κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα εδώ. Πολύ σημαντική λοιπόν επαναλαμβάνω ενίσχυση και εναρμόνιση της ε, εθνικής νομοθεσίας έτσι ώστε η πώληση αυτών των έργων τέχνης να εμποδιστεί, να υπάρχει απαραίτητα υποχρέωση πιστοποιητικών ενίσχυση της ποινική δίωξης, των κυρώσεων, της ε, διακρατικής ε, συνεργασίας σε επίπεδο αστυνομικών αρχών, δικαστικών αρχών. Η Ιντερπολ και η UNESCO πολλές φορές έχουν μεγάλη δυσκολία για να φτάσουν μέχρι τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πληρέστατος ο κατάλογος των στοιχείων μας δώσατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πανώνε της Criminal Intelligence Office της Interpol σχετικά με κοιμήλια τέχνης και πολιτικής εκλογίας που έχουν κλαπεί και στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτήν την δημόσια κρόαση και που καλέσατε την Interpol εδώ μου ζητήθηκε να παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών. Εάν όμως μετά έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και στις αρχές επιβολής νόμου στον τομέα αυτό, θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Πολιτισμικά αγαθά λοιπόν και παράνομη διακίνηση. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει λοιπόν ε, αυτά τα αγαθά. Τα εγκλήματα τώρα που έχουν, να, έχουν σχέση με αυτά έχουν διασυνδέσεις με ε, οργανωμένο έγκλημα και ε, αποτελούν μεγάλη απειλή είναι ένα διεθνές φαινόμενο και χρειάζεται αποτελεσματική πολιτική με μέτρα τα οποία θα ληφθούν σε διεθνές επίπεδο. Για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό με ε, επιθυμητά αποτελέσματα, η Interpol έχει δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για τα έργα τέχνης η οποία ε, εμπλουτίζεται συνεχώς και την οποία συμβουλευόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ύπαρξή της. Καταρχάς είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να προστατεύσουμε κάτι το οποίο δεν ε, γνωρίζουμε. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση της διακίνησης, παράνομης διακίνησης αγαθών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες να έχουν μία πλήρη βάση δεδομένων των πολιτισμικών τους αγαθών και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν σε περίπτωση κλοπής ή εξαφάνισης κάποιου πολιτισμικού αγαθού έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ ε, ο Διεθνής Μηχανισμός Αναζήτησης και ανα... εντοπισμού και ανάκτησης του αγαθού αυτού. Επίσης, χρειάζεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών η οποία θα βελτιώσει την, ε, το έργο μας και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης τόνισε την ε, σημασία της καταπολέμησης παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών. Το 2008 μάλιστα στηρίχθηκαν οι δράσει τη Interpol για την βελτίωση και τον εμπλουτισμό τη βάση δεδομένων και τη συμπερίληψη ενός συστήματο αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα από τα ίδια τα κράτη-μέλη και θα χρησιμοποιεί τις νεότερες τεχνολογίες, για παράδειγμα ε, ταυτοποίηση των διάφορων εικόνων κτλ αποφασίστηκε το 1995 να δημιουργηθεί μία αρχικό ε, ομάδα εργασίας. Αυτή η ομάδα αποτελούταν από εμπειρογνώμονες της ε, αστυνομίας από εννέα διαφορετικές χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Το 2009 και το 2010 Είχαν λάβει χώρα πολλές ενημερωτικές συνεδριάσεις και ως αποτέλεσμα οδηγηθήκαμε σε τρεις επιθανές λύσεις έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί βάση δεδομένων της Interpol. Θα δείτε στην οθόνη τη δυνατότητα που έχει κάποιος να ζητήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας μετά του δίνεται ένας κωδικός σε χρήστη με τον οποίο μπορεί να μπει στη βάση δεδομένων και να αναζητήσει κάποιο αντικείμενο. Στις 17 Οκτωβρίου 2011, ως αποτέλεσμα αυτών, η Ιταλία αφιέρωσε ένα τμήμα της ε, Ιταλικής αστυνομίας στο πρόγραμμα αυτό, τον εξυγχρονισμό δηλαδή της βάσης δεδομένων της ε, Ίντερπολ. Αυτό έγινε υπό το πρόγραμμα ΙΣΑΚ. Δεκαπέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό ως ε, συνδικαιούχοι. Και ο Γενικό Γραμματέας της Ιντερπολ έχει επίσης συμπεριληφθεί ως εταίρος και συνεργάτης. Το πρόγραμμα αυτό, το, το ΣΑΚΙ, ολοκληρω, θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, 27 Αυγούστου 2015. Και οι δράσεις που αναπτύσσει έχουν να κάνουν με την εφαρμογή ενός συστήματος ενημέρωσης και μηνυμάτων στην βάση δεδομένων της Interpol που θα διευκολύνει την εισαγωγή και καταγραφή πληροφοριών. Η δεύτερη δράση του προγράμματος είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών που θα μεταδίδουν άμεσα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων του κάθε κράτους μέλους. Όπως είπε και η κυρία Κώστα προλίγου, Τις δύο λοιπόν βάσεις δεδομένων της ε, Interpol. Θα έχουν όλα τα κράτη-μέλη την, δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να, αυτή τη βάση δεδομένων και να την συμπληρώνουν επίσης. Έπειτα, τρίτη δράση, η ενσωμάτωση ενός εργαλείου συγκριτικής αναζήτησης για τον εντοπισμό των ε, αντικειμένων. Και τέταρτη δράση, ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος, ε, διάφορα προγράμματα κατάρτισης των αστυνομικών αρχών που θα ε, ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές για το πώς θα χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο απαιτεί μια ε, πολυσχεδή προσέγγιση, όχι μόνο τον, ε, στη συμμετοχή των ε, αστυνομικών αρχών, αλλά και των αρχών που διαχειρίζονται πολιτισμικά αγαθά. Ο καθένας έχει το δικό του συγκεκριμένο ρόλο και συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο για να γίνει πιο εύκολη η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ε, πολιτισμικά αγαθά που έχουν κλαπεί ή εξαφανιστεί, όλοι οι φορείς, τα μουσεία, οι διεθνείς οργανισμοί, οι έμποροι έργων τέχνης, οι εμπειρογνώμονες κτλ. συγκεντρώθηκαν και οδήγησαν στη δημιουργία της βάσης δεδομένων της Interpol το 2009. Αυτή η βάση δεδομένων τώρα είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί να την συμβουλευτεί. Να αναζητήσει αντικείμενα και σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή βασιλεμένο, ένα πολύ καλό εργαλείο αναζήτηση. Σα παροτρύνω να την επισκεφτείτε και να δείτε μόνοι σα με τα μάτια σα το τι έχουμε καταφέρει. Μετά τον Αύγουστο του 2015 θα αλλάξει η εμφάνιση της κυρίας Ελίζας της βάσης δεδομένων της Ίντερπολ. Έχουμε μία νέα επιφάνεια εργασίας εξυγχρονισμένη και απλουστευμένη. Θα είναι λοιπόν πιο εύκολο να ψάξει κάποιος και να αναζητήσει ένα αντικείμενο στη βάση δεδομένων. Αυτά ενημερωτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αυτό το πρόγραμμα Psyche μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για ένα κοινό σύστημα τήρησης ε, τράπεζα δεδομένων. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Ε, παρακαλώ να μείνετε εντός των δύο λεπτών Σδρογεύσκη, Γραμματικάκης ε, και οι υπόλοιποι ομιλητέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε αυτές τι πληροφορίε Και έχω και μια ερώτηση για τον κύριο Πανώνε. είχαμε πληροφορίες ότι 36.000 αντικείμενα σε 120 χώρες τα αναζητεί η Ιντερπολ και ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου στο Υπουργείο Παιδείας είχαμε κάποιες δράσεις σχετικά με την ε, αναζήτηση και ανάκτηση αυτών των αντικείμενων. Πάνω από 8.000 εργατέχνης μεγάλων δημιουργών, Renoir και λοιπόν, θα πρέπει βεβαίω να δούμε και την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Μεταξύ άλλων μέσω ε, οίκων δημοπρασίας. Ο κύριος Γραμματικάκης παρακαλώ. Εγώ θα αρχίσω κυρία Πρόεδρε από μια εμπειρία που εσείς αναφέρατε τη διαδρομή δηλαδή της Επιτροπής Πολιτισμού από την Αφίπολη στη Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να πω ότι χάρη και σε εσά ε, αυτή η διαδρομή είχε φοβερή επιτυχία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το συνδέω με την ερώτησή μου. Ε, οι εκλεκτοί σημερινοί ομιλητές καλύπτουν το θέμα αυτό του, αν θέλετε, της παράνομης λαθρεμπορίας από τρεις πλευρές, από την νομική, από την πλευρά της UNESCO και πολύ καλή έκπληξη για μένα από την μεριά της Interpol που φαίνεται μάλιστα να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ γνωστό θέμα ωστόσο, θα το αναφέρω, παλιό αλλά πάντοτε εχμηρό που είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα που αγγίζει και τους τρεις ε, αξιόλογους ομιλητές. Όπως ίσως ξέρουν πολλοί από εσά, τα μισά περίπου γλυπτά του Παρθενώνα αφαιρέθηκαν βία από το ναό επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία, πουλήθηκαν στο Βρετανικό Σημείο από τον Λόρδο Έλβιν, Έλγιν και άρχισαν οι προσπάθειες για την επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα. Είμαι, είμαι πάρα πολύ ήπιος για το θέμα. Ε, το κύριο επιχείρημα για την άρνηση του Βρετανικού Μουσείου να παραχωρήσει σε κάποιο ελληνικό μουσείο την κυριότητα των γλυπτών του Παρθενώνα ήταν η έλλειψη κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και τη συντήρησή τους. Από το 2009 όμως και εύχομαι σε όλους σας να επισκεφθείτε το νέο λαμπρό μουσείο της Ακρόπολης που προκαλεί πράγματι αλλά και τη θλίψη των επισκεπτών για την ορατή καταστροφή ή και την απουσία πολλών αγαλμάτων. Ε, βέβαια η αναγκαιότητα της επιστροφής των γλυπτών έχει επιβεβαιωθεί και από την επίσημη θέση, το ξέρετε, τη UNESCO με βάση την αρχή της διατήρησης της ακαιρεότητας των μνημείων, της ακαιρεότητας το υπογραμμίζω, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το Βρετανικό Μουσείο πρόσφατα απέρριψε την πρόταση του UNESCO να διαδραματίσει ένα ρόλο μεσολαβητή ε, για να ε. επιτευχθεί κάποιο είδους αν θέλετε άμεση ή μακροχρόνια λύση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και τους τρεις ομιλητές, ίσως είναι και θέμα Ιντερπόλ, αλλά ειδικά τον κύριο Ρενό και τον κύριο Μπλαχέ, ποια είναι η στάση τους σχετικά με αυτό το ζήτημα πέραν από κάθε φανατισμό και να με συμβουλεύσετε μένα με ποια μέτρα και ποιες κινήσεις η Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια επίλυση του σπουδαίου του θέματος που βέβαια κυρία Πρόεδρος θα αποτελέσει και ένα πολύ καλό οδηγό για το μέλλον που σήμερα μας απασχολεί. E ε, η κυρία Τρούπελ και, με, και μετά θα κλείσουμε με την τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση όλων των μελών του πάνελ. Κατενόησα ότι γίνονται προσπάθειες συνεργασίες, αλλά μεταξύ των οργανισμών σας θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο καλύτερης συνεργασίας, αποτελεσματικότερης συνεργασίας, ένας, ένας καλύτερου συντονισμού μεταξύ αυτών των τραπεζών δεδομένων για την καλύτερη καταγραφή του τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη λαθρεμπορία. Μήπως έχετε μεγέθη για, την, για το συνολικό μέγεθος του φαινομένου. Δηλαδή πόσα εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έργα τέχνης ή κοιμήλια ε, ιστορικής πολιτιστικής αξίας. Ποια δηλαδή είναι και μίλια ιστορικης πολιτιστικης αξιας ποια δηλαδη ειναι η προοδος ε, που έχουμε σημειώσει στην ταυτοποίησή του και τι δουλειά μας μένει ακόμα να κάνουμε για να τα ταυτοποιήσουμε όλα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σβέντροβα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες του βήματος για τις παρουσιάσεις τους και για την εμπειρία που εδώ μας μετέδωσαν σήμερα. Εγώ ήθελα να θέσω το ερώτημα στον κύριο Πανώνε. Η καταπολέμηση κατά του παράνομου, μάλλον η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ιστορικών και πολιτιστικής αξίας κοιμηλίων είναι πάντοτε ένα δύσκολο εγχείρημα. Φαντάζομαι ότι έχετε σημειώσει κάποιες επιτυχίες στην καταπολέμησή σας αυτή Έχουμε κάποιες καταχωρήσεις σε αυτά τα μητρώα στα οποία αναφερθήκατε στους καταλόγους. Αλλά έχουμε και παραδείγματα αφαίρεσης από τους καταλόγους αυτούς. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα μητρώα για να ταυτοποιήσουμε τους κατόχους, τους παράνομους κατόχους αυτών των αγαθών. και τελικά στην προσπάθειά μας αυτή τα καταφέρνουμε, είμαστε αποτελεσματικοί, δηλαδή έχετε μεγέθη σχετικά με την παράνομη διακίνηση, κυκλοφορία ή ποσοτικά στοιχεία για τον κατάλογο αυτό και συνολικά για τα κοιμήλια που είναι αντικείμενο κλοπής Ίσως να εννοεί η ομιλήτρια. Ε, να απαντήσω στα Ιταλικά λέει ο μιλητής χάριν πρακτικότητους. Δεν μιλάμε για 20, χρόνες, 20 χώρες και χιλιάδες αντικείμενα. Μιλάμε για εκατομμύρια αντικείμενα που κυκλοφορούν παρανόμως από αυτά που έχουν κλαπεί αν θέλουμε να τα πιστοποιήσουμε και να καταγράφονται αυτά σε μητρώα σε όλες τις χώρες θα πρέπει να καταγράψουμε όλα εκείνα που είναι αντικείμενα παράνομης εξκαφής που παρουσιάζονται ακόμα και σε μουσεία τα οποία όμως δεν έχουν καταχωριστεί νομίμως όλα αυτά τα αντικείμενα όπως έλεγα από παράνομη εξκαφή που μετά παρουσιάζονται ενδεχομένως σε προσωρινά σε προσωρινές εγκαταστάσεις παράνομα υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία αγαθών και αντικειμένων μιλούμε για χειρόγραφα για αγαλματίδια για απεικονίσεις ε, τα οποία κλέβονται μερικές φορές από μουσεία και διατίθενται παράνομα στο εμπόριο Και επομένω για να απαντήσω και σε μια άλλη πτυχή της ερώτησής σας, προκειμένου να ποσοτικοποιήσει κανείς το ποσοστό, αν θέλετε, της επιτυχίας μας, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο επιχείρημα γιατί δεν ξέρουμε καν το συνολικό αριθμό των ερευνών που διεξάγονται. Επίσης, όπως πάντα προσπαθούμε να θυμίσουμε, και εγώ τουλάχιστον πάντα το κάνω, μία έρευνα αστυνομικής αρχής είναι αντίστοιχη όπως για οποιαδήποτε άλλο πεδίο δικαίου ή κώδικα. Και εγώ πολύ συχνά γι' αυτό κλείνω τις παρουσιάσεις μου με τα λόγια που βλέπετε στη διαφάνεια. Δηλαδή, το καθήκον της αστυνομικής αρχής είναι να ταυτοποιήσει τους δράστες και τα αντικείμενα και να προσπαθήσει να έχει επαρκείς πληροφορίες και ενδείξεις ώστε να φέρει τους δράστες αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα των κλαπέντων αγαθών πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ότι πολύ συχνά είναι προϊόντα τα οποία διατίθενται και σε νόμιμο εμπόριο. Υπάρχει δηλαδή νόμιμο εμπόριο πολιτιστικών στοιχείων. Το που δύσκολο είναι να καθορίσει κανείς και να πιστοποιήσει την παράνομη προέλευσή τους και άρα εισαγωγή τους στο κύκλωμα του νομίμου εμπορίου. Εγώ παλαιότερα είχα ειδίκευση ε, στα θέματα της καταπολέμησης της αστυνομικής αρχής και πολύ συχνά είχαμε προβλήματα με την υλοποίηση την εφαρμογή της οδηγίας 97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι για την επιστροφή ενός αντικειμένου θα έπρεπε να πιστοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία της εξόδου από τη χώρα προέλευσής τους και το χώρο παράνομης εξκαφής, το οποίο ήταν αδύνατον. Γιατί θα έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας ε, επιστημονικής μελέτης και έρευνας και για πολλά από αυτά τα αντικείμενα δεν θα δικαιολογεί το κάνει το κόστος μια τέτοια μελέτης και πλήρεστατης έρευνας. Κάτι λέει η πρόεδρος εκτός μικροφώνου, δεν την ακούσαμε. Οπότε και για την εφαρμογή και τη λύση των συνθήκων και συμβάσεων, εφόσον μια χώρα προσυπογράφει μια, τη σύμβαση για παράδειγμα της UNESCO του 70, αλλά μετά δεν εφαρμόζει τη δική της νομοθεσία, τις δικές της εθνικές διατάξεις και δεν δημιουργεί συγκεκριμένη μονάδα διώξεως της αστυνομικής αρχής για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας της παράνο, του παράνομου εμπορίου στοιχείων τέχνης και πολιτικής κληρονομιάς, η όλη προσπάθεια είναι πολύ πιο δύσκολη. Εξού και για την ερώτησή σας σχετικά με τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των αρχών των συναρμοδίων. Οι αστυνομικές αρχές, ναι, υφίστανται και δραστηριοποιούνται. Αλλά ε, ο περιορισμός είναι ότι και οι αστυνομικέ αρχές δεν μπορούν παρά να δραστηριοποιούνται και να δρουν επί τη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Άρα έναντι του παράνομου εμπορίου έργων τέχνης ή στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ακριβώς η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των εθνικών πλαισίων νομοθεσία. Υπάρχουν εγκλήματα κατά της παγκοσμίας ε, πολιτιστικής ε, ανθρωπότητας σε μία χώρα που σε άλλη χώρα δεν ορίζονται ως τέτοια. Και επομένω η συνεργασία των αστυνομικών αρχών υπό την έννοια αυτή περιορίζεται και είναι αναποτελεσματική. Ακόμα και αν είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, πρέπει να σα διακόψω, λέει ο Πρόεδρος, διότι δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος ε, Πλό. Πολύ σύντομα. Όσον αφορά τον υπολογισμό και των ε, αντικειμένων αυτών, αλλά και ποια είναι η αξία τους, δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία. Πρόκειται για λαθρεμπόριο, για παράνομες ε, εμπορικές κινήσεις. Φυσικά και έχουμε σήμερα εικόνες δορυφόρου από τις τοποθεσίες της ε, Παλμύρας και αλλού βλέπουμε φυσικά αντικείμενα σπασμένα ή όχι και αυτό που σήμερα ξέρω είναι ότι όλα αυτά έχουν ε, φύγει, έχουν πουληθεί και βρίσκονται κυρίως ιδιωτικές ε, συλλογές. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την αξία αυτών των ε, έργων τέχνης. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από τις αστυνομίες της Συρίας, του Λιβάνου, της Τουρκίας. Πρόκειται για αντικείμενα τα οποία τελικά κατασχέθηκαν μετά από αστυνομικές έρευνες είτε στα σύνορα και σήμερα προστατεύονται σε κάποιους ασφαλείς χώρους στη Συρία. Η Τουρκία επίσης διαθέτει σήμερα πολλά αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Το θέμα των ε, μαρμάρων του Παρθενώνα, των ε, συζητήσεων που γίνονται, όπως ξέρετε υπάρχει μια επιτροπή που στην UNESCO ασχολείται με το θέμα αυτό και πρόκειται για τα αντικείμενα αυτά τα οποία έχουν βγει από την Ελλάδα πριν από το 1979. Πρόκειται για αντικείμενα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αυτής της Επιτροπής και η Γενική Διευθύντρια της UNESCO η οποία έχει κάνει έτοιμα για διαμεσολάβηση και αυτή η αίτηση έχει μέχρι τώρα μείνει αναπάντητη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επαναλαμβάνω πρόκειται για μία αίτηση η οποία αυτή τη στιγμή εξετάζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει όμως αντιδράσει προς το παρόν για το θέμα αυτό. Μια και μιλούμε για συμφωνία, ίσως καλό θα ήταν να βρούμε και κάποια άλλη στοιχεία, μπας και μπορέσουμε να τη σκεφτούμε ως συμφωνία και λειτουργήσει. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, σχετικά με, την, ε, με αυτά που υπόθηκαν από τα μέλη, εγώ πιστεύω ότι η κεντρική έννοια είναι η συνεργασία. Δηλαδή, να παρατηρήσει κανείς πώς ε, συνεργάζεται η Ένωση με την UNESCO και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και μην ξεχνούμε τις τελωνιακές αρχές, τους τελωνιακούς ελέγχους, γιατί ακριβώς αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της μετάβασης. Και έχουμε και πρόσφατα παράδειγμα επιτυχούς παρέμβασης των τελωνιακών αρχών. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε την πτυχή αυτή. Και για να κλείσω με το εμβληματικό θέμα των αναγλήφων του Παρθενώνος, όπως είπε και ο κ. Πλόνσο, ε, πρόκειται για ευαίσθητο θέμα γιατί αφορά θέμα που προηγείται των θεμελιωδών νομικών κειμένων που χρησιμοποιούμε σήμερα και για χώρα που ευρίσκεται υποκατοχή, εν πάση περιπτώσει είναι αντικείμενο διεθνούς διπλωματίας και διαπραγματεύσεων. Υπάρχει μια επιτροπή διακυβερνητική, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες συνεννόησης και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε, εν πάση περιπτώσει, μια λύση πρωτότυπη θα έλεγα ή αυθεντική γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε τελικά μια διέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες λέει η Πρόεδρος για το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό απόγευμα γεμάτο από τόσες πολλές ιδέες που μπορούν να μας εμπνεύσουν. Τώρα θα έλεγα να προβάλλουμε τώρα αυτό το βίντεο του κυρίου Μαχμούν Αμπτούλ Καρίμ που είναι υπεύθυνο ε, από το Μουσείο το Αρχαιολογικό της Συρίας ε, θα είναι μόνο στα αγγλικά, δεν μπορούσαμε να το διερμηνεύσουμε αυτό. Παρακαλώ φορέσετε ε, τα ακουστικά διότι είναι ο ήχος λίγο χαμηλός όπως μου λένε. Παρακαλώ. Good morning. Many ancient Syrian cities have been subject to damage and destruction and some castles and archaeological buildings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 Ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο αυτό, την πολύ σημαντική αυτή μαρτυρία. Διότι ο καθηγητής που μας μιλούσε εδώ ήταν πραγματικός μάρτυρας των γεγονότων αυτών μαζί με τους σπουδαστές του. Έχουμε ακούσει ξανά και ξανά τις εκκλήσεις του ε, για βοήθεια από την ε, διεθνή κοινότητα υποστήριξη και προστασία σε, όχι μόνο των μουσείων και των πεδίων αρχαιολογικής ε, εξκαφής αλλά γενικώ της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, ξέρω ότι και η Λουξεμβουργιανή Προεδρία και ο Υπουργός ε, Πολιτισμού που θα συναντήσουμε αύριο έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα του πολιτισμού αλλά γενικώ όλοι μας έχουμε την ευθύνη να δώσουμε απτές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα ελέγχθησαν σήμερα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες. Ε, έχω την εντύπωση τώρα, ή μάλλον δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει κάτι να προσθέσει εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, η κυρία Σακητάνη, η κυρία Γκαρκόβα, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει κάτι να προσθέσει, κάτι να πει. Απλώς εγώ ήθελα να εξασφαλίσω το εξή, επειδή γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή εργάζεται επί του θέματος των εισαγωγών δηλαδή της οδηγίας μας λείπει για τις ε, εισαγωγικούς ελέγχους και προς την υποστήριξη όλων αυτών των συνεργατικών ε, προσπαθειών μαζί με την UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι στα σκαριά και νομίζω ότι και η Κομισιόν προετοιμάζει μια ανακοίνωση για την πολιτιστική διπλωματία όπως λέγεται. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια προκαταρχική ενημέρωση από αυτού. Ευχαριστώ. Oui, Ευχαριστώ πολύ. Σα καλωσορίζω όλους εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, για αυτήν την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την Επιτροπή Πολιτισμού και το Κοινοβούλιο για την πολύ σημαντική οθέτηση ψηφίσματος και της έκθεσης μάλιστα του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο. Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, χαρακτηρίζεται ως έγκλημα και φυσικά σήμερα ξέρουμε ότι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές χρησιμοποιείται και σαν μέσο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Φυσικά δεν υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Χρειάζεται δράση νομική, αστυνομική, τελωνιακή, αναπτυξιακή εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες, διπλωματική δράση, εξωτερική πολιτική. Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι φορείς και η Επιτροπή πρέπει να συνεισφέρουν. Τι κάνουμε εμείς στην Επιτροπή. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει κανονισμούς για την απαγόρευση εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών από το Ιράκ και από τη Συρία. Πρόκειται για κάτι που έχει προχωρήσει, υπάρχουν ήδη πρώτες κατασχέσεις έργων τέχνης ε, που προέρχονται από τις χώρες αυτές. Καταπολεμούμε επίσης, σαν μέρος του οργανωμένου εγκλήματος, αυτή την παράνομη διακίνηση μέσω της Ίντερπολ και πολύ συγκεκριμένα έχουμε χρηματοδοτήσει την σύσταση του Διεθνούς ε, Παρατηρητήριου για την ε, παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών που διαχειρίζεται το ΙΡΚΟΜ και ο κύριος Φλώσσα και άλλοι αναφέρθηκαν στο σχέδιο που χρηματοδοτούμε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στη Συρία για κατεπίγουσες δράσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με την UNESCO, το ΙΡΚΟΜ και παρακολουθούμε βεβαίως ε, τις τελευταίες εξελίξεις στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Επίσης, στην Επιτροπή το 2011 προετοιμάσαμε μία έρευνα για την παράνομη διακίνηση στο λαθρεμπόριο των πολιτιστικών αγαθών και το Συμβούλιο Τζάι έχει ζητήσει βεβαίω από όλα τα κράτη-μέλη την κύρωση της σύμβασης της UNESCO το 1970. Τώρα, ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που έχουμε αναλάβει και μελλοντικέ δράσεις. Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, που υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να ληφθούν μέτρα για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και θα ξεκινήσουμε και μια νέα μελέτη για το παράνομο εμπόριο και την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτιστικών αυτών αντικειμένων. Αυτό στα πλαίσια του προγράμματος 2015-2018 για τον πολιτισμό θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμά μας και ελπίζω ότι μέσω αυτής της μελέτης θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν πιο ε, ενημερωμένο απολογισμό αυτού που συμβαίνει στον τομέα αυτό και ε, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε υιοθετώντα ε, μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να προτείνουμε κάποια τέτοια μέτρα. Θέλουμε βεβαίως να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με την UNESCO. Σήμερα το πρωί και με τον κύριο Πλόνς συναντηθήκαμε, εκπρόσωποι πολλών υπηρεσιών της Επιτροπής, για να εξετάσουμε και να εμβαθύνουμε την περαιτέρω συνεργασία μας και να ε, δημιουργήσουμε μια πολύπτυχη απάντηση, αντιμετώπιση για να καταπολεμήσουμε αυτήν την μάστιγα της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών. Σας ευχαριστώ για τις σημαντικές αυτές ε, πληροφορίες. Ε, νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο θα έχουμε και πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Αρκετά στοιχεία από αυτά που αναφέρατε χρειάζονται ενδελεχέστερη εξέταση και με την υποστήριξη της Επιτροπής και αναφέρομαι κυρίως ε, στο θέμα της ε, επιστροφής των αντικειμένων αυτών και μιας, ενός επιχειρηματικού πλαισίου ενισχυμένου στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή. Και έχω την εντύπωση ότι από τους νομικούς του Διεθνούς Δικαστηρίου ε, ε, για τα όσα είπαν σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας νομίζω ότι έχουμε συγκεκριμένες επιπτώσεις οικονομικές αντίκτυπο και αναφέρθηκε και ο καθηγητής νωρίτερα πολύ συγκεκριμένα για τις ε, εντός οικών αντιφατικές πολεμικές υποστηρίξεις ή προσπάθειες υποστήριξης αλλά από τη στιγμή για την οποία ε, οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποστηρίζουν συγκεκριμένε δράσει επί του εδάφου, αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μια στήριξη και εκπαιδευτική και ε, πιο συγκεκριμένη δηλαδή βοήθειες. Και νομίζω ότι κάπω έτσι προέκυψε και η ανάγκη του να προχωρήσουμε στην διεύρυνση αυτού του προγράμματο ΣΑΙΚΙ και να έχουμε την κοινή χρήση και συνεργασία επί τη βάση αυτής της ε, κοινή τράπεζα δεδομένων. Και όπως είπε και ο κύριος ε, Πλόνς, ε, την ενίσχυση των διατάξεων του ποινικού κώδικα των χωρών και της σωστή υλοποίησης και εκτέλεση των διατάξεων αυτών. Προφανώς θα συζητηθούν και σε άλλα βήματα διάφορα στοιχεία που συζητήθηκαν από διάφορους και συζητούνται και στη δική μας τη χώρα, τη δική μου. Δηλαδή για την διεύρυνση <clears throat> των καθηγόντων των αρμοδιοτήτων των κυανοκράνων του ΟΗΕ σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις και προς την υπεράσπιση στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. και νομίζω ότι ε, σε σχέση με αυτά που είπαμε η γενοκτονία υπό την έννοια της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κάτι που μπορεί να συμπεριληφθεί στην εντολή και τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο αρμοδιότητων του ΟΗΕ. Να κλείσω απλώς λέγοντας, αναφέροντας κάτι που δεν αφορά μόνο στην Ιταλία ότι δεν τελειώνει εδώ ο διεθνής διάλογος και η Διεθνή ε, συνεργασία. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στην έξπο του Μιλάνο ο Υπουργός Πολιτισμού Φραντσισκίνη έχει καλέσει όλες ε, τις χώρες που εκπροσωπούνται ε, ή στην ΕΞΠΟ και τους οργανισμούς που είναι πάρα πολλοί. Έχουμε ζητήσει και από την κυρία Μπούκοβα ε, εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και καλοδεχούμενοι όλοι οι άλλοι που θα θέλουν να συμμετάσχουν. Ένα βήμα, ένα ενιαίο βήμα ώστε να επανακινήσουμε ζωηρά την προστάτη αυτή προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις χώρες μεταξύ των οποίων και τις χώρες εκείνε που δεν έχουν συνυπογράψει, δεν έχουν επικυρώσει την σύμβαση. Και νομίζω ότι είναι σωστά όλα αυτά που λέμε από τον περασμένο Μάρτιο για να δεσμευτούμε και να ενεργοποιηθούμε από το θέμα αυτό. Ευχαριστώ όλους ε, τους εμπειρογνώμονες, τα αξιότιμα μέλη του πάνελ, παρακολουθούμε ενδιαφέρον το έργο σα. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά για να επανέλθουμε. Με αυτό θα κλείσουμε τώρα, γιατί έχουμε μετά μέσω του συντονιστέ. παρακαλώ.